Liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Ο κύριος Επίτροπος έχει έρθει ήδη και επομένω θα είναι ο Σονούπο μαζί μας. Σας ε, χαιρετίζω όλους και μπορούμε να ξεκινήσουμε ήδη με τα σημεία 1 και 2. Μπορούμε να τα κλείσουμε πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει για την ημέρα διάταξη, αν έχετε προτάσεις για τροποποίηση, εάν όχι, που να θεωρήσουμε ότι τις έχουμε εγκρίνει. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις τώρα από τον Πρόεδρο και ήθελα την προσοχή σας στο σημείο αυτό. Καταρχήν, για την επιτροπολογία, για τις λεγόμενες κατευθυντικές γραμμές ATC. Ο κύριος Ρούμπι, αλλά όχι μόνο, είχε, διατυπώσει μια αντίρρηση για τη διαδικασία αυτή της επιτροπολογίας, οπότε θα πρέπει να επιληθούμε το θέμα τους αυτού μαζί με τους ε, συντονιστές. Εάν λοιπόν, αν μπορέσουμε να βρούμε ένα δρόμο να προχωρήσουμε, θα σας αναφέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο στόχος μας είναι στις 4 Μαΐου στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας να εγκρίνουμε το αντίστοιχο ψήφισμα. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να σας πω. Δεύτερον, στη συνεδρίασή μας Τετάρτη και 5η Μαΐου θα καθυστερήσει λίγο <clears throat> η έναρξη της συνεδρίασής μας γιατί η κυρία Κρούζ η οποία θα ερχόταν ε, στις 4 Μαΐου είχε αναβάλει την προηγούμενη της την παρουσία της θα την αναβάλει και πάλι. Επομένως το πρώτο σημείο θα, δεν θα αντιμετωπιστεί και θα πρέπει να ξεκινήσουμε στις 10 η ώρα το πρωί αντί στις 9, οπότε μπορείτε να κάνετε και ένα δεύτερο πρωινό. Αυτό δεν είναι τόσο δυσάρεστο. Και κατά τη διάρκεια του πρωινού μπορούμε και να συζητήσουμε αν θέλετε. Τρίτη παρατήρηση, λόγω της κατάστασης που δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο, δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε μια πρόσθετη συνεδρίαση. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να τύχουν ψηφοφορίες. Και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση, θα ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση στις 8.45 λίγο νωρίτερα από τις άλλες συνεδριάσεις μας. 11 Μαΐου, 8 και 45 λοιπόν είναι η πρόσθετη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να εξασφαλίσουν οι πολιτικές ομάδες να είναι αρκετοί τουλάχιστον από κάθε πολιτική ομάδα ώστε να έχουμε απαρτία. 8 και 45 έως 9 και 15 στις 11 Μαΐου θα γίνει η ψηφοφορία για την οδηγία που αφορά τα κτίρια και κάτι άλλο δεν θυμάμαι. Τα δύο σημεία που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στο Στρασβούργο και δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Πέντε λεφτά θα κάνει η ψηφοφορία, όχι περισσότερο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να φέρουμε στο, στην Ολομέλεια αυτό το θέμα και γι' αυτό έχουμε πίεση χρόνου. Τρίτο σημείο στην ημέρησια διάταξη και μετά θα σταματήσω. Είναι τα θέματα της έγκρισης των πρακτικών της 22-23 Φεβρουαρίου, 1 Φεβρουαρίου και 22-23 Μαρτίου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ε, αίτηση να αλλάξουν τα πρακτικά. Εάν όχι, θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά αυτά. Και το σημείο 3 έχει και αυτό αντιμετωπιστεί. Και τώρα έχουμε στο σημείο 4 και ε, <clears throat> θα πρέπει να κλείσουμε όλες αυτές τις επαφές με τους επιτρόπους για να μπορούμε να έχουμε κλείσει όλες αυτές τις επαφές με τους επιτρόπους προτού συζητήσουμε για το νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν και είχαμε αποφασίσει πρώτα να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις και μετά να συζητήσουμε. Στην Ολομέλα δεν ξέρω αν αυτό είναι απόλυτα ευφυές. Και θέλουμε πάντως να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους επιτρόπους για να ξέρουμε ποια είναι και η άποψή μας σε σχέση με το πρόγραμμα της Κομισιόν. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν κάποιες προτάσεις και από τη δική σας πλευρά για την αντίδραση που θα έχουμε προς την Κομισιόν. Χθε συναντηθήκαμε με το Γενικό Διευθυντή ΛΟ σε σχέση με το σχέδιο δράσης και υπήρξαν διάφορες απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν γιατί η Κομισιόν με αυτό το οποίο <clears throat> προέβλεπε έχει καθυστερήσει και θα έχουμε αυτά τα στοιχεία αργότερα σε σχέση με το πρόγραμμά της. Ο κύριος Λό είπε ότι εάν θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε μια ενδιάμεση έκθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι πλήρως έτοιμο το πρόγραμμά μας. Η προσωπική μου λοιπόν άποψη δεν έχει νόημα να ζητήσουμε μια προσωρινή έκθεση η οποία δεν έχει κανένα δεσμευτική, κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα Ας δεχτούμε ότι θα γίνει αργότερα η πρόταση της Κομισιόν, αλλά είναι μια ουσιαστική πρόταση για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Για... Νομίζω ότι αυτό είναι πιο λογικό, πιο οικονομικό από πλευράς χρόνου και θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μια σωστή ανάλυση του προγράμματος της Κομισιόν και να πάρουμε μια εμπεριστατωμένη θέση για αυτά. Αυτή ήταν η τελευταία πληροφορία που ήθελα να σας ε, δώσω και τώρα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα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 Μα έχουμε το πρόβλημα αυτό με τον Επίτροπο, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε την, την ψηφοφορία στις 10. Ίσως. Θα ήταν χρήσιμο να ήταν λίγο πιο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει θα δώσω το λόγο στους διάφορους ε, συναδέλφους. Χολ, Βίνκνερ και κάποιος άλλος. Κύριε Σόντι, Είναι πρώτη πρώτοι που θα θέσουν ερωτήματα στον κύριο Επίτροπο. Αυτό είναι αξιόλογο που ξέρετε ήδη θα ρωτήσετε. Τη στιγμή που δεν έχει πει τίποτα ο Επίτροπος ακόμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα εγκάρδια τον Επίτροπο Ταγιάννη. Είναι ο πρώτος Επίτροπος ο οποίος έρχεται ενώπιόν μας για να μας παρουσιάσει το τμήμα που τον αφορά σε σχέση με το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα γιατί στις 10 πρέπει να ψηφίσουμε. Επομένω δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, θα δώσω αμέσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Ταγιάννη και μετά θα ακολουθήσουμε οι παρατηρήσει και οι ερωτήσει. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά ήρθα με τα πόδια γιατί υπάρχει μια διαδήλωση η οποία έχει προκαλέσει κάποια προβλήματα κυκλοφορίας. Ας περάσουμε αμέσως στα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και να κάνω και μια ανακοίνωση για μια απόφαση που πήρε η Επιτροπή σήμερα το πρωί γύρω από έναν πολύ σημαντικό τομέα, τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπως γνωρίζετε είναι μεγάλη χαρά για μένα και το εννοώ αυτό να επιστρέφω στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή έχω περάσει 15 χρόνια σε αυτές τις αίθουσες ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, της πολιτικής μου ζωής και κάθε φορά που επιστρέφω εδώ είμαι ιδιαίτερος ευτυχής γιατί έχω τη δυνατότητα να συναντήσω πάρα πολλούς συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα. Να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω σήμερα στα πλαίσια του διαλόγου του διοργανικού το νομοθετικό πρόγραμμα το οποίο υιοθέτησε στις 4 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο περιλαμβάνει απαριθμοί τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα επιμείνω και στα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου μου και τη δική σας Επιτροπή. και θα κλείσω με την ανακοίνωση για <clears throat> τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκινούμενα οχήματα, την οποία κυκλοφόρησε ή αποφάσισε μάλλον ε, στην τελική της φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 η ώρα σήμερα το πρωί. Θα σας την παρουσιάσω δηλαδή την ανακοίνωση πριν τη δώσουμε στον τύπο. Ποιες ήταν οι στρατηγικές πρωτοβουλίες μας. Εμείς όπως είδατε <clears throat> μέσω μέσα στα έγγραφά μας στοχεύουμε να υπάρξει μια νέα πολιτική στον τομέα της βιομηχανίας για μια αηφόρο ε, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μια ανταγωνιστική και πολυπίκυλη βιομηχανική βάση. Η νέα αυτή βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, οριζόντια, καινοτόμος και αηφόρος να δίνει κίνητρα για τη δημιουργικότητα, να αναπτύσσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να λειτουργεί στρατηγικά σε σχέση με τις πρώτες ύλε. Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συνοδεύει τις ε, ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά εμείς δεν μπορούμε σαν δημόσια διοίκηση να αντικαταστήσουμε τη σωστή διαχείριση των επιχειρήσεων. Αλλά παρόλα αυτά θα συνοδεύσουμε τις αλλαγές και θα προσδώσουμε ανταγωνιστικά στοιχεία στο βιομηχανικό μας δίχτυ. Προβλέπουμε ένα ολόκληρο σύστημα για την σωστή και ισόρροπη λειτουργία της αγοράς που δίδει νομικές βεβαιότητες στους οικονομικούς εταίρους. Η Ευρώπη έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός Απλά δεν έχουμε ακόμα την δυνατότητα να συντονίσουμε στο βαθμό που θέλαμε και να καταστήσουμε αλληλέγγυη την οικονομική μας δραστηριότητα. Υπάρχει ανάγκη προς την κατεύθυνση αυτή. Κάποιες βιομηχανίες όπως η αυτοκίνητο βιομηχανία <coughs> θα πρέπει να επανειδρυθούν σε εισαγωγικά και αυτό το λέγει άλλωστε και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οικοαποτελεσματικά αυτοκίνητα σήμερα από το πρωί. Ο πρόεδρος Μπαρόζο αποφάσισε στα πλαίσια αυτής της πολιτικής να δημιουργήσει μια ομάδα επιτρόπων που να ασχολούνται με τον συγκεκριμένο τομέα. Εγώ θα είμαι ο συντονιστής έτσι ώστε να συζητήσουμε σε πολιτικό επίπεδο τις συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση αυτή επί τη βάση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς και των ελλείψεων που χαρακτηρίζουν κάθε τομέα. Η αδίποτε πρόταση από πλευρά σας <clears throat> θα γίνει καλοδεχούμενη και ελπίζω να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε εκ νέου τα θέματα αυτά και στο Στρασβούργο όταν εσείς πιστέψετε ή θεωρήσετε ότι θα πρέπει να συναντηθούμε. Μία πρώτη εισφορά θέλετε ήταν η θεωρησετε οτι θα πρεπει να συναντηθουμε μια πρωτη σφορα θελετε ηταν η διασκεψη για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας που οργανώθηκε στο κτίριο Σαρλεμάνια και Δευτέρα, προχθές. Πήραν μέρος πάρα πολύ σημαντικοί ομιλητές και φυσικά ήταν και ο πρόεδρος <coughs> της Επιτροπής σας, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή του σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Ήταν και ο συνάδελφος Αλμούνια, ήταν ο προεδρεύων Σεμπαστιάν και τα λοιπά. Η δεύτερη στρατηγική πρόταση αφορά το πρόγραμμα δράσης για την έρευνα και την καινοτομία. Η υποστήριξη στην καινοτομία είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής μας στον τομέα της, της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Συνεργάζομαι με την Γιόγκαν Κουίν έτσι ώστε να μπορέσουμε το φθινόπωρο να καταθέσουμε μια νέα πρόταση βασιζόμαστε σε μια ερμηνεία της έννοιας της καινοτομίας που περιλαμβάνει όχι μόνο ερευνητές αλλά χρήστες, βιομηχανία, ε, κατασκευαστές και γενικότερα το κοινό. Η καινοτομία πρέπει να παίξει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας και γι' αυτό προετοιμάζουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καινοτομούν Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του προγράμματος δράσης. Η δημιουργία ευρωπαϊκού ε, χώρου ε, soluzioni innovative per il servizio pubblico europeo, in particolare incoraggiando gli acquisti pubblici. ενός ευρωπαϊκού χώρου επιχειρηματικού κινδύνου, όπως επίσης και ενός χώρου ε, γενικά καινοτόμων πρωτοβουλειών. Θα υπάρξει επίσης και ε, αναθεώρηση της πολιτικής μας ε, για τα διάφορα επίπεδα ποιότητας τα οποία στοχεύουμε και θα υπάρξει συγκεκριμένη δράση έτσι ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μπορέσει να κυριαρχήσει και ε, με μια πολιτική σύγχρονη για τα διάφορα επίπεδα ποιότητας τα οποία μπορεί να εξάγει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στις λεγόμενες αναδυόμενες αγορές. Οι άλλες πρωτοβουλίες μας αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, ανάλογα με το κράτος μέλος, έχουν διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας. Σε κάποιες χώρες υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάκαμψης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, κάνει έναν κατάλογο, θα έλεγα, των βημάτων προόδου στα οποία ε, προέβησαν οι διάφορες χώρες. Η διάσκεψη για το λεγόμενο Small Business Act που προβλέπεται στη Μαδρίτη τέλος Μαΐου αρχές Ιουνίου. αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Θα απευθύνω έκκληση προς το Κοινοβούλιο έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει συμφωνία σε κρίσιμα νομοθετικά μέσα σχετικά με την εφαρμογή του Small Business Act. Αναφέρομαι στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών από αυτό εξαρτάται κατά πολύ η δημιουργία ενός περιβάλλοντος πολύ πιο κατάλληλου για την εύρυθμη λειτουργία των μικρομεσαίων. Έχει περάσει 1,5 χρόνος από τις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακόμα φαίνεται ότι στο Συμβούλιο δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Καλό λοιπόν το Κοινοβούλιο να, συνεισφέρει και αυτό με κάποιες θετικές προτάσεις γιατί αν δεν φτάσουμε σε μια ανάγνωση, <clears throat> σε μια λύση στη πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης, σημαίνει ότι θα χάσουμε ένα επιπλέον χρόνο. Και σε μια τόσο ευαίσθητη φάση της οικονομικής κρίσης κάτι τέτοιο είναι πολυτέλεια και πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να καταλήξουμε. Ένα άλλο θέμα είναι το Εράσμους για τους επιχειρηματίες. Είναι μια πρωτοβουλία στην οποία εγώ ενδιαφέρομαι για την οποία ιδιαίτερα περιορισμένου μεγέθους αλλά μπορεί να αναπτυχθεί. Από το 2009, ε, το 2009 έγιναν 90 ανταλλαγές επιχειρηματιών και προετοιμάζονται άλλες 90 για φέτος και έχουν κατατεθεί άνω των 2.000 υποψηφιωτήτων από πλευράς των, του επιχειρηματικού κόσμου. Το πρόγραμμα Έρασμους για τους επιχειρηματίες θα μετατραπεί σε μόνιμο πρόγραμμα σε δύο χρόνια και τότε θα αποκτήσει τη σωστή του διάσταση. Τώρα για το διάστημα και η διαστημική πολιτική είναι βασική και για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Η συνθήκη της Λισαβόνας προσδίδει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και είναι η νομική βάση για την μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρώπης στην έρευνα για το διάστημα. Οι υπηρεσίες μου εργάζονται για τη διαμόρφωση μίας ανακοίνωσης για τη διαστημική πολιτική για να διευκρινιστούν οι μελλοντικέ δραστηριότητες της Ένωσης προ την κατεύθυνση αυτή. Η υιοθέτηση αυτή της ανακοίνωση προβλέπεται να γίνει το Σεπτέμβριο. Παράλληλα θα παρουσιαστούν την άνοιξη του 2011 προτάσεις νομοθετικές για το μελλοντικό διαστημικό πρόγραμμα έτσι ώστε ε, να τα λάβουμε υπόψη μας και για το επόμενο χρηματοοικονομικό πλαίσιο 2014-2020. Σε σχέση με τον Γαλιλαίο GMS έχουμε ήδη διαμορφώσει κάποια σημεία υπεροχής. Για να υπάρξει επιτυχία <clears throat> του προγράμματος αυτού θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει την κατάλληλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είδα, ε, ε, ε, είπα ήδη στην ακρόασή μου εδώ και λίγους μήνες. Δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να υιοθετήσουμε αποφάσεις για τις μελλοντικές προκλήσεις και τους προσανατολισμούς μας, αν πρώτα δεν έχουμε ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά τις απόψεις του Κοινοβουλίου για να αποφασίσουμε τι πράγματι θέλουμε να κάνουμε μαζί, από κοινού. Πριν λοιπόν καταλήξουμε στην ανακοίνηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος Γκαλιλαίο, θα πρέπει να συζητήσουμε μέχρι το καλοκαίρι τα θέματα αυτά αναλυτικά. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές επιλογές που θα πρέπει να γίνουν για το μέλλον του Γκαλιλαίου και πρόθεσή μου είναι να ξεκινήσουμε εκ νέου το θέμα της σωστής λειτουργίας του διοργανικού πάνελ του Γκαλιλαίου έτσι ώστε να καταστεί ένας κατεξοχήν χώρος πολιτικού διαλόγου και ανταλλαγής πολιτικών εμπιστευτικών πληροφοριών γύρω από τη λειτουργία του Γκαλιλαίου. Είναι ένα πάνελ το οποίο έχει εργαστεί μέχρι τώρα, αλλά μπορεί να εργαστεί καλύτερα και να συντονίσει καλύτερα τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες άλλωστε πήραν την εντολή από μένα να συνεργαθούν στενά και με τις δικές σας υπηρεσίες και με τις υπηρεσίες του Συμβουλίου, για να μελετήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες βελτίωσης του Γκαλιλαίου. Ένα άλλο θέμα σημαντικό, πολύ σημαντικό, αφορά τις πρώτες ύλε. Είναι ένα στρατηγικό πολιτικό θέμα για την οικονομία της Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται φυσικά από τις εισαγωγές των πρώτων ύλων ε, για τα μετάλλα και ορυκτά, σαν παράδειγμα. <clears throat> Όπως ακριβώς συνέβη και το 2 και πιο πρόσφατα στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020, Υιοθετήσαμε τους βασικούς προσανατολισμούς της ανακοίνωσής μας για τις πρώτες ύλες, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, πρόσβαση σε πρώτες ύλες στο εσωτερικό της Ένωσης. Δεύτερον, πρόσβαση σε πρώτες ύλες εκτός Ένωσης. Και τρίτον, αποτελεσματική χρήση και ανακύκλωση πρώτων ύλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανακοίνωση πριν από το τέλο του χρόνου, έτσι ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική ανάλυση για την πρόσβαση στι πρώτε ύλε στα πλαίσια τη οικονομική συγκυρία και των προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να, υπάρξει, να υπάρξουν εγγυήσει για την αηφόρο ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή οικονομία. Τον Ιούνιο θα πάω στην Άντισα Μπέμπα και θα συζητήσουμε με τους Αφρικανούς εταίρους το θέμα αυτό. Οι πολιετής προοπτικές. Ε, τώρα στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας μου, ίσως μακρηγορώ λίγο, ζητώ συγγνώμη, αλλά καλό θα ήταν να σας ενημερώσω για ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι κάνουμε αρκετά πράγματα και γι' αυτό ακριβώς αναγκάζομαι να ομιλώ ιδιαίτερα. Το πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα. Είμαι ικανοποιημένος. Παρά την περιορισμένη χρηματοδότηση καταφέραμε να φτάσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλαμε. Έχουμε τώρα αρχίσει την προπαρασκευή για τον επόμενο κύκλο βασιζόμενοι στα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Τώρα κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Είμαι απολύτως πεπισμένος για την μεγάλη στρατηγική και πολιτική σημασία που έχει το δίκτυο αυτό και τις θετικές επιπτώσεις που έχει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στις επιχειρήσεις και στο οικονομικό μας σύστημα εξαρτάται από την οικονομική από την κοινωνική αντίληψη των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο έχει επιβαρυνθεί μέσω της οικονομικής κρίσης. Έχουμε πετύχει ήδη αρκετά αποτελέσματα τους πρώτους μήνες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το REACH. Το REACH θα συνεχίσει να είναι μια βασική μου προτεραιότητα και θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε να στεφθεί από επιτυχία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν σεβαστεί το πρώτο χρονικό όριο για την εγγραφή τους για την επόμενη χρονική περίοδο διάρκειας μάλλον του ΡΙΤΣ. Αν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Σύμφωνα με τις ανηλυμένες υποχρεώσεις οι οποίες ακούστηκαν νομίζω και στην ακρόαση που οργανώσατε πρόσφατα, θα καταλήξουμε σε πρακτικές προσπάθειες έτσι ώστε να βοηθήσουμε την βιομηχανία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη λειτουργία της ομάδας επαφής των διευθυντών που διευκολύνει τις ευθύνε που έχουν αναλάβει οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες. Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αδειοδοτήσεις και τα δικαιώματα, χαίρομαι για τη συμφωνία στην οποία κατέληξα με τον Επίτροπο Ποτότσνικ και που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της μικτής μας επίσκεψης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών στο Ελσίνκι, ε, και νομίζω ότι το ταχύτερο δυνατόν θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. Ο οδηγός για την αδειοδότηση, ο κατάλογος των ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται θα κυκλοφορήσουν έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η απαιτούμενη νομική ασφάλεια που είναι θα έλεγα χρήσιμη και προαπαιτούμενο για την πρόοδό στον τομέα και αυτό θα ξεμπλοκάρει και τη διαδικασία αδειοδότησης δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταθέτουν τις αιτήσει τους και να προασπίζονται την ύπαρξη και αδειοδότηση συγκεκριμένων ουσιών τη απουσία εναλλακτικών. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάποια στοιχεία γύρω από την απόφαση την οποία υιοθετήσαμε με γραπτή διαδικασία σήμερα το πρωί μια διαδικασία η οποία αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα καθαρά και οικοαποτελεσματικά αυτοκίνητα. Όλες οι παρεμβάσεις αυτές ε, θα προσδώσουν αξία θα έλεγα στο παραγωγικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σεβόμενη και την αρχή της επικουρικότητας κρινοθετικότητα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σαν παράδειγμα βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής σε πολλά κράτη-μέλη, Γαλλία, Ισπανία, Δανία, Πορτογαλία. Και υπάρχει ε, η προοπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να υιοθετήσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει στην απανθρακοποίηση σε εισαγωγικά της βιομηχανικής παραγωγής και θα προωθήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες ε, για τις νέες τεχνολογίες ε, υπολογίζοντας να χρησιμοποιήσουμε το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και βελτιώνοντας γενικά ε, την βιοαποτελεσματικότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση. Νομίζω ότι θα ληφθούν πολλές πρωτοβουλίες, θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω κάποιες από αυτές. Πρώτον, οικονομικά κίνητρα, υποστήριξη στην καινοτομία των αηφόρων μορφών ενέργειας, καθορισμός στόχων του Κοινωνικού Ταμείου από τον επόμενο χρόνο ε, για να ενθαρρύνουμε την λειτουργία του, ρυθμίσεις για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των αυτοκινητουμένων οχημάτων, και επίσης υπάρχουν και μέτρα ειδικά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι εξίσου ασφαλή με τα συμβατικά. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε κάποια κοινά standards που αφορούν το σύνολο ε, των οχημάτων τα οποία φορτίζουν ηλεκτρικά και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι ε, προσβατά από το κοινό. Συγκεκριμένα επίπεδα λοιπόν παραγωγής, οικονομικά κίνητρα και στήριξη της έρευνας στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιούμενες εθνικές προτάσεις και λύσεις εδώ. Πρέπει να συνεργαστούμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι μια στρατηγική την οποία θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογείτε ήδη από σήμερα, γιατί θυμίζω σήμερα το πρωί, πρωί έχει δύο κατευθύνσεις, βελτιώσεις των μηχανών εσωτερικής καύσης για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου και βελτίωση των κινήτρων που μπορεί να δοθούν για την παραγωγή ηλεκτρικών κινητήρων, κινητήρων κινουμένων με βιοκαύσιμα και με υδρογόνο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια συνεργασίας και στα πλαίσια της περίπτωσης 21. Εν πάση περιπτώσει η ανακοίνωση σήμερα το πρωί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι νομίζω ένα κομβικό σημείο που αποδεικνύει την αιμονή μας ε, στα θέματα τα οποία είχαμε πει ότι θα ακολουθήσουμε στη φάση που ζήτησα την εμπιστοσύνη σας πριν έξι μήνες δηλαδή. Μακρηγόρησα το ομολογώ, αλλά σας ευχαριστώ για την θερμή σας υποδοχή και είμαι στην διάθεσή σας για να δώσω πιθανώς απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα χρόνου που σας είπα ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 10 ε, αλλά έχω πάνω από 10 ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν νομίζω θα προλάβουμε όλοι. Εκτός, εάν θέλετε, ε, εκτός αν μπορείτε να περιοριστείτε σε ενός λεπτού ερώτηση μονάχα. Εγώ σας πρότεινα να το κάνουμε αυτό έτσι να προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε την προσοχή σας μονάχα στο ερώτημα, αφήστε τη αυροφροσύνη, τα ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά τον Επίτροπο, μας ξέρει και αυτό πολύ καλά, να εστιάσουμε την προσοχή μας στα ερωτήματα και ίσως θα προλάβουμε μέχρι τις 10. Ξεκινάμε λοιπόν. κύριο κύριος Βίνκλα έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για την έρευνα και την καινοτομία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η καινοτομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως και θα ήθελα να ξέρω στα πλαίσια της προετοιμασίας αυτού του σχεδίου για την καινοτομία αν υπάρξει λοιπόν κάποια σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την έρευνα και την καινοτομία άκουσα ότι θα υπάρξει μια ομάδα κρούσεως, μια task force για τα θέματα αυτά. Θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη συνολική αυτή προβληματική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Επίτροπε, Πώς σχολιάζετε τον αντίκτυπο των τελευταίων εξελίξεων στι παγκόσμιε διαπραγματεύσεις για τη χρήση του άνθρακα σε σχέση με την ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, και θα μετακυληθεί αυτό στο κόστος παραγωγής, αν όχι, πώς ακριβώς ε, ε, θα κινηθούμε στα πλαίσια της βιομηχανικής μας πολιτικής, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον κλάδο, αλλά για να μην έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Δεύτερον, ε, για τον ανταγωνισμό όλες οι μεγάλες χώρες ε, που στις μεγάλες συμβάσεις εισαγάγουν ρήτρες προτιμησιακές. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, πώς προβλέπετε να υπάρχει αμοιβαιότητα μέσα στις μεγάλες συμβάσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας στη διεθνή σκηνή. Δεν θα ήθελα να επιβαρύνω ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα πυκνό και μεγάλο. Χαίρομαι για τη φροντίδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καθίσταται πλέον βασικό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τον Επίτροπο να δώσει την προσοχή του, να στρέψει την προσοχή του και να φροντίσει κάποιες μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες ε, στη λειτουργία τους. Παρόλα αυτά απασχολούν σχεδόν 10 εκατομμύρια, 10 ε, εκατομμύρια εργαζομένους. Είναι εταιρείε οι οποίες παράγουν γενικά κέρδος αλλά δεν είναι όμως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις έχουν πολλές μορφές ε, ε, λειτουργίας όπως είναι εταιριστική κτλ. Κύριε Χολ, σύντομες ερωτήσεις. Ε, πρώτον, στην τυποποίηση για τα ηλεκτρικά οχήματα θα μεριμνήσετε ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε και τις ευφυείς τεχνολογίες ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε και για αποθήκευση ηλεκτρισμού τα οχήματα δεύτερον για το Γαλιλαίο. Συμφωνώ ε, ότι πλέον δεν είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, ούτε καν βιώσιμο είναι τεχνολογικός πώς ε, για τις υποδομές μας. Οπότε τι είδους ανάλυση ωφέλους θα κάνετε για να συγκρίνετε τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με άλλα προγράμματα υποδομών όπως το ε, Super Grid στη Βόρεια Θάλασσα ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο και για την βιομηχανική υποστήριξη, παραδείγματο χάρη, για την μεταρρύθμιση του βιομηχανικού κλάδου σχετικά με την ε, τροποποίηση των ε, σιδηροδρομικών δικτύων. Κάνετε τέτοιες αναλύσεις πάλι για τον Γαλιλαίο. Ε, είπατε ότι η Κίνα δεν έχει απελευθερώσει το φάσμα και άρα υπάρχει σύγκρουση για το Γαλιλαίο. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και τέλος, οι πρώτες ύλες η πρόσβαση εκτός Ευρώπης είναι ένα θέμα διακυβέρνησης επίσης και άρα θα πρέπει οι εξορρυκτικές βιομηχανίες να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια ε, ε, για να μην ε, αυξηθεί η διαφθορά. Δηλαδή είναι θέμα συνοχής στην πολιτική μας εφόσον γενικότερα θέλουμε να βελτιώσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση εκτός Ευρώπης. Η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το επιχειρήν για το, το έρασμος για τους επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα πρόβλημα ανεργίας μεταξύ των νέων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μεγαλώσει αυτό το πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι έχουμε μονάχα 2 εκατομμύρια για το 2010-2011, είναι πολύ λίγα λεφτά <clears throat> και στα προγράμματα αυτά δεν λαμβάνει υπόψη η παροχή υπηρεσιών από τους επιχειρηματίες. Επίσης, είναι σημαντικό να είναι τεχνολογικά ουδέτερη η πρόταση για τα, για τα εναλλακτικά αυτοκίνητα και να συνεχίσουμε και την έρευνά μας στις μηχανές εσωτερικής καύσης και όχι μονάχα στα ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κύριος Φράγκο. Επίτροπε, θα ήθελα να ξέρω τι προτίθεστε να κάνετε για να βελτιώσετε την διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις ε, συμπραξίες κοινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς θα τις ενθαρρύνετε να δραστηριοποιούνται μέσα από την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία υποστήριξη. Επίσης, πώς θα στηρίξετε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης για τη Μεσόγειο. Ε, κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις και μία ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ η καλή πρωτοβουλία σας για τα πράσινα αυτοκίνητα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά να δούμε γενικά ποιε είναι οι άλλε εναλλακτικέ λύσει, δηλαδή να ακολουθήσει ένα τεχνολογικά ουδέτερο δρόμο η, τεχνο, η Κομισιόν στα τεχνολογικά θέματα και επίση πώ βλέπετε τι πρωτοβουλίε αυτέ σε σχέση με τι πρωτοβουλίε άλλων περιοχών του κόσμου. Οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι επενδύουν μαζικά για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις, ε, τη βιομηχανία αυτή εναλλακτικών αυτοκινήτων. Επίση, ένα ερώτημα θα υπάρξουν ευρωπαϊκά μέσα, ευρωπαϊκά κονδύλια για την πρωτοβουλία των πρασίνων αυτοκινήτων που θα προκαλέσουν περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την ε, ε, καινοτομία. Δεύτερη παρατήρηση, η έρευνα που προσανατολίζεται προς την καινοτομία. Το έθεσε αυτό το θέμα ο κύριος Βίνκλερ, ίσως θα πρέπει να συνοηθείτε και με την αρμόδια επίτροπο για τα ερευνητικά θέματα, ώστε να μην υπάρξει μονάχα γενική εστίαση, αλλά μια ιδιαίτερη εστίαση στα θέματα καινοτομία που πρέπει στο κέντρο αυτών των προσπαθειών. Λινέκ, πρώτον, ε, Έχουμε δέκ προσώπου από πολιτικέ ομάδε ε, που συμμετείχαν στι διαπραγματεύσει ε, για το σχέδιο ανάκαμψη οικονομία. Θα τηρήσετε τι υποσχέσει σα στην Επιτροπή για αυτό το σχέδιο ανάκαμψη οικονομία. Διαπραγματευτήκαμε επίση το σχέδιο ΣΕΤ ε, μας έλειπε χρηματοδότηση και μας λείπει ακόμη. Το 50% λείπει. Θα τηρήσετε τις υποσχέσεις σας γι' αυτό. Και τρίτον, πότε μπορούμε να προβλέψουμε κοινά πρότυπα για τις ε, μπρίζες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά την Ευρώπη. Ριέρα Μαρουγέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι η Κομισιόν θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μία ουδέτερη τεχνολογικά προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία, τεχνολογία ηλεκτρικής κίνησης αυτοκινητών είναι πολύ πιο προθυμένη. Οι κατασκευαστές έχουν ήδη παρουσιάσει μια πλειάδα μοντέλων και σύντομα θα υπάρχει εμπορία αυτών των μοντέλων σε μεγάλη κλίμακα. Μήπως θεωρείτε ότι θα πρέπει να δώσουμε μια ταχύτερη μια μεγαλύτερη προώθηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να χρησιμοποιηθούν στην Ευρώπη πριν από άλλε καθαρέ τεχνολογίε. Επίση, ένα άλλο ερώτημα, η καινοτομία είναι φυσικά παράγον ανταγωνιστικότητα τη επιχειρήση, αλλά υπάρχει και ένα άλλο παράγον, τον οποίο δεν έχουμε αναφέρει αρκετά και αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χειροτομήσουν, αλλά τα προϊόντα και οι διαργασίες τους θα πρέπει να απευθύνονται σε μια ευρύτερη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς την διεθνοποίηση των διαδικασιών και των προϊόντων. Πώς θα προωθήσει η Κομισιόν αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Μπίτικοφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι κύριε Επίτροπε που σε σχέση με την πολιτική προτύπων ε, έχετε συζητήσει με τους Αμερικανούς εταίρους μας Προηγουμένως ήταν ο Επίτροπος Φερχόγγεν υπεύθυνο για τα θέματα αυτά, για το Διατλαντικό Συμβούλιο Επιχειρηματικότητος. Αυτά τα θέματα τώρα έχουν περάσει σε εσά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς επίσης <clears throat> να δώσετε την πρέπουσα προσοχή για το θέμα των προτύπων τα οποία πρέπει να θεσπίσουμε από κοινού και θα με ενδιέφερε να ακούσω από εσά ποιες είναι οι προτεραιότητες οι οποίες κατά την άποψή σας έχουν να κάνουν με την πολιτική προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα πρέπει να μεταφερθούν στο διατλαντικό διάλογο. Επίσης έχετε αναφερθεί στο Small Business Act και εδώ πέρα θα πρέπει να σταθούμε και στο θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών. Εγώ θέλω να επιχειρηματολογήσω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικές ομάδες αυτού του Κοινοβουλίου, αλλά είναι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, <clears throat> οι οποίες πιέζουν πάρα πολύ ώστε αυτή η οδηγία να αναφέρεται και στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Ο κύριος Έντσο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάτι τον <coughs> Επίτροπο. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει κονδύλια για να ενθαρρύνει τις online συναλλαγές, ε, κυρίως ε, ε, για τους ανέργους μέσα από ένα νέο χρηματοπιστωτικό μέσο που θεσπίστηκε στις 8 Μαρτίου. Θα χρησιμοποιήσετε αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο. Κάτι άλλο Ε, δεδομένη της διάσκεψης υψηλού επίπεδου που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, ε, εδόθησαν ε, κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, αντλήσατε κάποια συγκεκριμένα διδάγματα. Ο κύριος Παντά. Στην στρατηγική 2020 η χαμηλή χρήση άνθρακα και ενεργειακός αποδοτική οικονομία έχουν μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Ταυτόχρονα, αν δείτε τι έγινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2010 και κάνετε τη σύγκριση, δεν βλέπω αυτά τα θέματα να είναι ε, προτεραιότητες. Πώς το σχολιάζετε αυτό. Ο κύριος Βαλών, Βαλεών. Κυρία Βαλεών, ευχαριστώ για το θέμα των ε, πρώτων υλών. Αυτή τη στιγμή Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο η Κομισιόν έχει μια συνολική άποψη σε σχέση με τους πόρους που έχουμε υπομορφή πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θέλετε να ενθαρρύνετε τις εξορρυκτικές βιομηχανίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερη δυσκολία στο να έχουν πρόσβαση σε περιοχές που προστατεύονται από περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την έκκληση του Κοινοβουλίου να υπάρξει μια απαγόρευση της χρήσης κυανιούχων ενώσεων στην εξόριξη χρυσού, κάτι το οποίο θα ψηφίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα ασφάλειας, έρευνα στην ασφάλεια με 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα τα οποία έχουμε περάσει στον προϋπολογισμό το, κοινο, το Συμβούλιο τα περιέκοψε τα ποσά αυτά, εμείς τα επανεφάραμε ε, εμείς ως Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε λοιπόν το μέλλον της έρευνας, θέλετε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ασφάλεια του διαδικτύου και θέλουν να έχουν ένα διάλογο για προτυποποίηση και κοινά πρότυπα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βλέπετε αυτή η προοπτική. Δεύτερον, υπήρξε πάντα μια κοινή άποψη στο Κοινοβούλιο ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να υποστηριχθούν, αλλά να υπάρχει μια διάκριση μεταξύ στρατιωτικής και μη στρατιωτικής έρευνας. Αλλά βλέπουμε ότι ξαφνικά αναδύεται το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα και αυτό ίσω είναι προπομπό στρατιωτική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε πρέπει να διατηρηθεί αυτή η διάκριση μεταξύ στρατιωτική και μη στρατιωτική ε, έρευνα καταρχήν και εάν πράγματι είναι έτσι, θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια παρουσία στρατιωτικών φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας στην έρευνα για την ασφάλεια του διαδικτύου. Κυρία Τικάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ είμαι, γιατί είδα ότι με ψάχνατε. Για να μην εκτοπιστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η βιομηχανική παραγωγή και το ίδιο και με τι θέσει απασχόλησης, πρέπει οπωσδήποτε να καινοτομήσουμε και να καταστήσουμε πιο οικολογική την παραγωγή μα. Επίσης ε, θα πρέπει να τηρήσουμε τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιώτο ε, και ό,τι έχει προβλεφθεί για την περίοδο μετά το Κιώτο. Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να εξυγχρονίσει τις βιομηχανικές μονάδες ε, σχετικά με την πρωτοβουλία για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που έχετε παραμείνει πιστοί στον χρόνο που σας είχε τεθεί και έχετε τώρα μετά τις ε, ερωτήσεις τη δυνατότητα να ακούσετε τις απαντήσεις του κυρίου Επιτρόπου μέσα σε 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σύντομα σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν Χωρίς να μπορώ βέβαια να μπω στο βάθος των συζητήσεων αυτών, θα μπορούσαμε τις συζητήσεις αυτές να τις κάνουμε ελεύθερα και με ησυχία στο Στρασβούργο, στην επόμενη συνάντησή μας. Είμαι στη διάθεσή σας γι' αυτό. Πάντως, και ο κύριος Φράνκο και ο κύριος Βίνκλε αναφέρθηκαν στο θέμα της πρόσβασης στην πίστοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ θα υποστηρίξω όλες τις πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε δάνεια των μικρομεσαίων. Αυτό θα το κάνω με νέα χρηματοδοτικά μέσα και μέσω της στενής συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τα σημερινά μέσα χρηματοδότησης έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά τους. Θα προσπαθήσουμε επίσης να διαμορφώσουμε και ένα αποτελεσματικό χώρο επιχειρηματικού κινδύνου, <clears throat> δημιουργώντας ένα διαβατήριο αν θέλετε, ε, σε κάποια ταμεία τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με καλύτερο τρόπο και με περισσότερες εγγυήσεις συναντήθηκα με τον κύριο Μεϊστάντ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ε, μπορέσαμε από κοινού να συζητήσουμε τις νέες δυνατότητες ε, για μετά το 2013. Στις 6 Μαρτίου οργάνωσα ένα φόρουμ για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ένα φόρουμ το οποίο αφορούσε την πρόσβασή τους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε γραφειοκρατικό επίπεδο. Συμμερίζομαι λοιπόν τις ανησυχίες ιδιαίτερα του κ. Βίγκλα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις, το συγκεκριμένες εννοώ το ταχύτερο δυνατόν. Από τότε που ήμουν επίτροπος για τις μεταφορές ξέρω τις δυσκολίες που υπήρχαν ε, τις γραφειοκρατικές για κάποια προγράμματα όπως το Μάρκο Πόλο, τα οποία δεν ήταν εύκολα προσβάσιμα στις ε, επιχειρήσεις αυτές. Και χθε άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ενημερώνουν πήρε κάποια μέτρα για την ε, γραφειοκρατική απλοποίηση, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία. Ο κύριος Οντί έθεσε ένα θέμα το οποίο έχει επανειλημμένα τεθεί και συζητήθηκε και στην ακρόαση την οποία οργάνωσε η συνάδελφός τη και συμπατριώτησά του. Εάν το ερώτημά σας είναι αν εγώ είμαι υπέρ του φόρου ή όχι, εγώ να σας πω ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει αποκλειστεί από τον κανονισμό ως έχει σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε αργότερα αν θα χρησιμοποιήσουμε ή όχι τη δυνατότητα αυτή, αλλά είμαστε ουδέτεροι σε σχέση με αυτό. Για την κυρία Τόγια. Η κυρία Τόγια ε, επιμένει στο συγκεκριμένο θέμα των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο και παρουσιάζει ενδιαφέρον και για κοινωνικούς λόγους, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και επιβεβαιώνω το ενδιαφέρον μου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές της ειδική μορφής επιχειρηματικότητας που έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό βάρος. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις μέχρι τις μικρομεσαίες θα είναι στο κέντρο των δραστηριοτήτων μου τα επόμενα χρόνια. Γύρω από το ερώτημα το οποίο έθεσε η κυρία Καρβάλιο. Δική μου επιθυμία, κυρία Καρβάλιο, είναι να μετατραπεί η προπαρασκευιστική φάση του Εράσμους για επιχειρηματίες σε μόνιμο λειτουργικό πρόγραμμα ο προϋπολογισμός και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Θα πρέπει λοιπόν οι πιστώσεις να επαναξεταστούν και προβλέπεται ότι θα γίνουν αυξήσεις από το 2012 να φτάσουμε τουλάχιστον στα 7 εκατομμύρια, το 13 8 εκατομμύρια, ενώ σήμερα είμαστε στα 5 εκατομμύρια. Έχουμε δηλαδή με ένα κάποιο ε, ε, μια θετική πορεία θα πρέπει να υπάρξουν ε, περισσότερες οικονομικές δυνατότητες στο μέλλον, γιατί νομίζω θα αποδεσμευθούμε και από τις υποχρεώσεις τις οποίες επιπλέον δημιουργεί η προπαρασκευαστική φάση στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα είναι μια δυνατότητα που δίνουμε στους επιχειρηματίες να μάθουν από τις επιχειρηματικές δράσεις συναδέλφων τους σε άλλες χώρες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, καλύτερα αυτοκίνητα. Είναι μια ερώτηση την οποία έθεσαν πολλοί κοινοβουλευτικοί. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάθε μία από τις ερωτήσεις του, <coughs> συγγνώμη, ξεχωριστά. Αλλά θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες πρώτος απαντήσεις. Κάποιοι από εσά ρώτησαν αν θέλουμε εμείς να δώσουμε προτεραιότητα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή να είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε ουδέτεροι. Έχει μεγάλη σημασία το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι η Ισπανική Προεδρία έχει καταστήσει την ηλεκτροκίνηση σημαία θα έλεγα της, της δραστηριότητάς στο κείμενο το οποίο υιοθετήσαμε σήμερα το πρωί υπάρχει χώρος μεγάλος για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και για το υδρογονοκίνητο και για τα αυτοκίνητα γενικά που χαρακτίζονται καθαρά. Είναι σωστές οι παρατηρήσεις λοιπόν που ακούστηκαν σχετικά με την ανάγκη κοινών υποδομών. Δεν μπορούμε εμεί τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια ανάπτυξη της αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ορισμένε χώρε. Ξέρετε ότι η Ρωσία και η Κίνα επενδύουν πάρα πολλά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ευρωπαϊκές επιχειρήσει, η Fiat σαν παράδειγμα που κατασκευάζει ε, το μοντέλο Cinquecento ηλεκτροκίνητο στις Ηνωμένε Πολιτείε και όχι στην Ευρώπη και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μαρκιόνε, είπε ότι η Fiat σκέφτεται να παράγει τα ηλεκτροκίνητα, μικρά αυτοκίνητά της και στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει θέμα υποδομών και κόστους. Είναι προφανές όμως ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείες επενδύουν πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερες δυνατότητες επιλογών να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή κινητήρων διαφορετικής φιλοσοφίας, όχι δηλαδή εσωτερικής καύσης, έχουμε δύο πυλώνες. Απ' τη μία έχουμε την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε στον τομέα των κινητήρων εσωτερικής καύσης για να μειώσουμε τις εκπομπές τους βραχυπρόθεσμα. Και από την άλλη έχουμε μια δεύτερη στρατηγική υπέρ αυτοκινήτων και κινητήρων που να μολύνουν λιγότερο υβριδικών, ηλεκτρικών, με υδρογόνο κτλ. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών την οποία θα πρέπει να αναλύσουμε. Για το Small Business Act Α, όχι πάντα υπάρχει θέμα με τις μπρίζες που θα χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εμείς ζητήσαμε από την υπηρεσία προτύπων να αναπτύξει μέσα στον επόμενο χρόνο ένα εναρμονισμένο κανόνα ευρωπαϊκό για τη φόρτιση και επαναφόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων έτσι ώστε η επαναφόρτισή τους να μπορεί να γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο όταν περνάει κανείς τα σύνορα. Ο κανόνας θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μας πριν από την μαζική παραγωγή τέτοιου είδους αυτοκινήτων και γι' αυτό καλό και τους βιομηχανικούς εμπλεκομένους παράγοντες να καταλήξουν στον καλύτερο ε, δυνατό κανόνα. per eh, Για τα ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με αυτά που ζήτησε ο κύριος Έχλερ, Νομίζω ότι η καινοτομία και η έρευνα είναι δύο από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και που οδηγούν στην καινοτομία. Η καινοτομία είναι θεμελιώδης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σύντομα προετοιμάζει μία ανακοίνωση για την καινοτομία. Όπως είπα συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Γκέγαν Κουίν. Ήδη συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες μας και και τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Κάποια τμήματα των προοπτικών αυτών θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αναδιατυπωθούν και να προβλέψουμε στις γραμμές του προϋπολογισμού κάποιες αλλαγές υπέρ της βιομηχανικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται στο κέντρο του εγγράφου Ευρώπη 2020. Πρέπει λοιπόν αυτές τις ανηλυμένες πολιτικές υποχρεώσεις να τις μετατρέψουμε σε πράξεις. Τότε μόνο η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει στη διάθεσή της ένα ανταγωνιστικό παραγωγικό βιομηχανικό σχήμα και τότε μόνο θα επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις μας να καινοτομούν. Η καινοτομία χωρίς την έρευνα δεν μπορεί να υπάρξει όμως και γι' αυτό βασικό κριτήριο τουλάχιστον σε επίπεδο αρχών, βούλησή μου είναι να είναι σε θέση ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να καλύψει τις ανάγκες της έρευνας καλύπτοντας τα υπάρχοντα κενά. Σχετικά με ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο υπογράμμισαν πολλοί συνάδελφοι και άπτεται των πρώτων υλών και της χρήσης των πρώτων υλών. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Πολλές βιομηχανίες άφησαν, θα έλεγα, κάποια μηνύματα ανησυχητικά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Εγώ συναντήθηκα με εκπροσώπους πολλών επιχειρηματικών κύκλων οι οποίοι μου εξέφασαν τις αμφιβολίες τους και τις ανησυχίες τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα με πραγματικότητες εξωευρωπαϊκές που για πάρα πολλές πρώτες ύλε χαρακτηρίζονται από μονοπωλιακά χαρακτηριστικά, από μονοπωλιακές καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Δευτέρας, που του φόρουμ αυτού, Ακούσαμε πολλά μηνύματα από το βιομηχανικό χώρο και συμφωνήσαμε όλοι για την σημασία που έχει φυσικά η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όπως μπορεί να τα επιβεβαιώσει και ο πρόεδρός σας από την συνεδρίαση της Δευτέρας μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εμπειρογνώμονες του βιομηχανικού τομέα οι οικονομολόγοι που ασχολούνται με τη βιομηχανία και τα λοιπά συμπίπτουν στην διαπίστωση ότι είναι θετική η στρατηγική Ευρώπη 2020. Το πέρασμα λοιπόν από ένα οικονομικό σύστημα το οποίο να βασίζεται αποκλειστικά σε υπηρεσίες και σε χρηματοπιστωτικά είναι κάτι το αρνητικό. Πρέπει να περάσουμε σε μια μορφή ανάπτυξης πιο ισορροπημένη που να δίνει χώρο και βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, στη βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακυρώσουμε τον τομέα των υπηρεσιών. Όχι, θα πρέπει απλά να έχουμε μια ισορροπημένη θα έλεγα αντίληψη για τα πράγματα έτσι ώστε να αποφύγουμε ζημίες προβλημάτων που προκαλούνται από προβλήματα οικονομικής αυστηρά φύσης ε, που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική διαδικασία και αναφέρομαι στη συγκυρία αυτών των ημερών. Σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει για τις πρώτες ύλες με τις τρίτες χώρες δεν σημείωσα τυχαία τη συνάντηση που θα έχουμε στην Άντις με την Αφρικανική Ένωση, γιατί αυτές είναι χώρες παραγωγής πρώτων υλών. Γι' αυτό λοιπόν και επιμένω και σας έχω ήδη ανακοινώσει ότι εγώ θα είμαι στην Άντις και θα θέσω τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ευρώπη οι Ευρωπαίοι έχουμε κάθε συμφέρον να αναπτύξουμε μια ουσιαστική πολιτική παρουσία στην Αφρική. Όχι μια νεοαπικιακή πολιτική παρουσία, αλλά μια αναπτυξιακή για την Αφρική πολιτική, μια πολιτική υπέρ της σταθερότητας της Υπήρου αυτής. Δεν θέλουμε να υπάρχουν αυτά τα επίπεδα διαφθοράς που σοβούν σε κάποιες από τις αφρικανικές χώρες. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και στις στρατηγικές βιομηχανίες βασιζόμενοι στην ποιότητα του know-how μας, της τεχνογνωσίας μας, της διαχειριστικής μας ικανότητας και γενικά της τεχνογνωσίας που εξάγουμε ε, στην Αφρική και βοηθάμε να εργάζονται οι Αφρικανοί. Αυτό είναι ένα πλαίσιο σημαντικό για τις πρώτες ύλε. Οι πρώτες ύλε είναι ενταγμένες σε ένα σωστό, θα έλεγα, πολιτικό πλαίσιο ανάπτυξης για την Αφρική. Εδώ και ένα χρόνο στην Άπολη της Ιταλίας έγινε ένα σεμινάριο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και την Αφρική και ένας εκπρόσωπος αφρικανικής χώρας μου είπε ότι θα πρέπει να εμπλακείτε περισσότερο στη δημιουργία ε, υποδομών στην Αφρική. Γιατί αν εσείς οικοδομήσετε στην Αφρική ε, ένα σιδηρόδρομο σαν παράδειγμα, θα είστε και οι πρώτοι που θα ξέρετε τι μπορεί κανείς να βγάλει από το υπέδαφος των περιοχών από όπου θα διέρχεται ο σιδηρόδρομος αυτός. Συνεπώς λοιπόν δεν θα πρέπει εμείς απλά να πηγαίνουμε στην Αφρική με βαλιτσάκια γεμάτα δολάρια αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε πολιτικές αναπτυξιακές δράσεις. Το θέμα αυτό των πρώτων υλών είναι κυρίαρχο, πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Ένα άλλο θέμα, το οποίο ανακοίνωσα και πριν λίγες μέρες, είναι η πρόταση για την κατάρτιση ενός καταλόγου σπάνιων πρώτων υλών, η υποεξάντληση πρώτων υλών. Θέλουμε επίσης να εργαστούμε και στα πλαίσια προγραμμάτων για την έβρεση ε, ουσιών αντικατάστασης ή πρώτων υλών αντικατάστασης και να ενισχύσουμε τις μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης της βιομηχανικής των πρώτων υλών και αυτό είναι κάτι που απασχολεί και αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξορρυκτικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκά επίπεδα αυτή τη φορά. Τώρα για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουτικόφα ο οποίος ε, έθεσε το ερώτημά του σαφέστατα είναι ένα θέμα που βρίσκεται υπό εξέταση, είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούνται οι συντονιστές. Έχουμε ήδη καταλήξει σε μια πρώτη συμβιβαστική συμφωνία. Σε ό,τι με αφορά θεωρώ ότι η συμβιβαστική αυτή συμφωνία ήταν αρκετά καλή. Έχει σημασία να εργαστούμε και από πλευρά Κοινοβουλίου με διπλωματικό τρόπο απέναντι στο Συμβούλιο για να έχουμε την δυνατότητα να πιέσουμε και να υπάρξει ένα τέγγραφο τελικά από πλευρά Συμβουλίου. <clears throat> Το Συμβούλιο πάνω κάτω έχει ήδη συμφωνήσει στο συμβιβαστικό ε, αυτό κείμενο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι κατά. Προφανώς αυτό το B2B θα πρέπει να είναι τμήμα της στρατηγικής μας, αλλά το καλύτερο είναι μερικές φορές εχθρός του καλού. Έχει σημασία να στείλουμε γρήγορα μηνύματα προς την κατεύθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν θέλουμε να καταλήξουμε στο τέλειο άμεσα τότε θα συναντήσουμε την αντίσταση πολλών κρατών μελών. Εγώ λοιπόν εργάζομαι και συνεργάζομαι και με πολλούς βουλευτές για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτη ανάγνωση έτσι ώστε και τα τρία όργανα να βοηθήσουν αυτήν την εποχή κρίσης της ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμένα λοιπόν η στρατηγική που προτείνεται μου κάνει, από την άλλη θα πρέπει οι λύσεις αυτές να λειτουργήσουν συμβιβαστικά. Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν μπορώ να σας στείλω και γραπτές απαντήσεις στους βουλευτές τους οποίους δεν έδωσα απάντηση ε, πλήρη σήμερα. Προφορικά είμαι στη διάθεσή σας για μελλοντικές συναντήσεις και για συναντήσεις ατομικές εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν παρόν. Δεύτερον που απαντήσατε πλήρως. Και τρίτον που μας δίνετε τις ε, πληροφορίε στην Επιτροπή μας προτού δημοσιευτεί η πρόταση τη Κομισιόν. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχιστεί η επωφελή συνεργασία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τις ψηφοφορίες επιτέλους. Äh, Ερχόμαστε στην ψηφοφορία. Ελπίζω ότι οι πολιτικές ομάδες έχουν μετρήσει ότι είναι μονάχο απαραίτητος και ο σωστός αριθμός βουλευτών εδώ και δεν χρειάζεται να κάνουμε τροποποιήσει στη συνέχεια. Στα αποτέλεσματα της ψηφοφορίας σας ευχαριστώ εξ αρχής. Πρώτη ψηφοφορία λοιπόν. Είναι η έκθεση της κυρίας Ποδηματά και θα ήθελε να κάνει μια εξήγηση προηγουμένως, σύντομη σας παρακαλώ, αλλά Παρακαλώ, να έχετε, το λόγο σύντομα κύριε Ποδηματά. Πρόεδρε, ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλου και κυρίως τους κοιόδους εισηγητέ, όσου συνέβαλαν στι συζητήσει και στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση τη οδηγία για την σήμανση των προϊόντων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργεια. Ήθελα να ζητήσω την προσοχή σα σε ένα σημείο, το οποίο υπογραμμίζω και στη γραπτή ε, αιτιολογική έκθεση που σας έχω στείλει, και αφορά στην τελική συμφωνία που επετεύθη σε ό,τι αφορά στο θέμα της σήμανσης. Γνωρίζετε ότι η συμφωνία προβλέπει maximum τρεις ενεργειακές τάξεις πάνω από το A, δηλαδή μέχρι A+++, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 και την αιτιολογική σκέψη 22. Προβλέπεται επίσης ρήτρα αναθεώρησης της οδηγίας το αργότερο το 2014. Συνεπώς, στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων, της σήμαση των προϊόντων, πέρα δηλαδή από την τάξη A+++, πριν από το 2014 και τη συνολική αναθεώρηση της οδηγίας, θεωρώ δεδομένο και αυτή είναι η ερμηνεία που συμφωνήθηκε προφορικά με την Επιτροπή κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι θα υπάρξει αναταξινόμηση των ενεργειακών τάξεων και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώσει στη διάρκεια της ψηφοφορίας της οδηγίας στην Ολομέλεια αυτή την ερμηνεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάση, αλλά σας παρακαλώ μην κάνουμε συζήτηση τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον ε, τριμερή διάλογο μας είπε προφορικός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως η ερμηνεία αυτή στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ποδηματά δεν θα παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ιδανική συμβαστική πρόταση και δεν ισχυρίζομαι βέβαια δεν εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο οι συγγητές. Οι πράσινοι πάντως θα ήθελαν μία γραπτή διαβεβαίωση της προφορικής αυτής ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λύση είναι ότι θα επιβεβαιώσει στην ολομέλεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την ερμηνεία και ήθελα να σας ενημερώσω απλώς υπό αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συμβαστική. Ο κύριος Πρίζα από την Κομισιόν. Πρόεδρε, αγαπητή συγγήτρια, επιβεβαιώνω φυσικά την ερμηνεία σας, ε, κύριε Αποδηματά. Αν χρειαστεί να αναθεωρήσουμε την ταξινόμηση ε, ε, πριν την αναθεώρηση, προς τα κάτω φυσικά θα γίνει. Θα δούμε ποιο τρόπο μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Με γρατή διαβεβαίωση στην Ολομέλεια. Θα δούμε τι είναι ευκολότερο δεν χρειάζεται απαραίτητα να γίνει στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω αν θα παρευρεθεί ο Επίτροπος Ότιγκερ. Θα διαβουλευτώ με τον Επίτροπο για να βρούμε το βέλτιστο τρόπο ώστε να καθησυχάσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι όντω αυτή είναι η μοναδική πιθανή ερμηνεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> Ήμουνα σε αυτόν τον τριγωνικό διάλογο και είχαμε συζητήσει πράγματι το θέμα αυτό. Μία ώρα κάτσαμε και φάγαμε μαζί και τα συζητήσαμε τα θέματα. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία τη έκθεση που αντιματά. Ποιο υπερψηφίζει, παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, πρέπει να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εντάξει. Το αποτέλεσμα είναι ομόφωνη έγκριση. Συγχαρητήρια. Επόμενη ψηφοφορία η έκθεση Τικάου και εδώ υπήρξε ε, υπάρχει μια ψηφοφορία μονάχα ηλεκτρονικά αρχίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία όχι, όχι δεν γίνεται θέλει θέλετε να λάβετε το λόγο, θέλετε να πείτε κάτι για όλα αυτά σας παρακαλώ δεν μπορούμε να κάνουμε και πάλι συζήτηση για κάθε έκθεση που ψηφίζουμε Αλλιώ πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τη μείωση των ρηπαντικών εκπομπών και της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και αυτό ιδίως για περιοχές που δεν καλύπτονται από την εμπορία εκπομπών. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν μια θέση στην πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, <clears throat> ναι, αρχή την ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί η κάρτα σας. Εντάξει, θα το λάβουμε υπόψη μας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «52-53 ψήφοι υπέρ, ομόφωνα δεκτή, συγχαρητήρια λοιπόν. Ερχόμαστε στην επόμενη έκθεση, την έκθεση Βίνκλα έχετε ένα κατάλογο ψηφοφοριών. Σε κάποιο σημείο έχουμε και μια προφορική τροποποίηση και εδώ χρειάζομαι τη βοήθειά σα. Λοιπόν, τροπολογία 18, Ριέρα Μαδουρέλ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21 υπέρ μου. 21 εκπίπτει. Προχωράμε και φτάνουμε στην ένα της εσωτερικής αγοράς. Υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 20 ποδηματά, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ίσως πρέπει να κάνουμε έλεγχο γιατί ήταν μικρή διαφορά. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για επαλήθευση. Κλείνει. Απορρίπτεται πράγματι. 22 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, ψήφι κατά, αποχές, δεκτή. Η 26 έχει εκπέσει, συμβαστή τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 31 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές <clears throat> απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 ψήφι υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ Η 47 έχει αποσυρθεί. Ξέχασα να το πω. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρι... Ε, εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή 68. 66 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, η 5 της ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχή δεκτή. ΙΜΚΟ 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή. <clears throat> Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 10 υπέρ κατά <clears throat> αποχές 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 εκπίπτει 81 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται συγγνώμη 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 με χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 97 καλύπτεται. 98 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές Απολύτω. 101 με προφορική τροποποίηση. Παρακαλώ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 102 ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, ναι, γίνεται δεκτή πράγματι. <coughs> Συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος. 100, 102 ήταν αυτή. 103 έχει εκπέσει. 104 υπέρ. 104 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 105 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 106 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 107 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 108 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή αιτιολογικές σκέψεις, 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή, 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή, 15. Έχουμε μια προφορική τροπολογία από την κυρία Ριέρα Μαδουρέο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μερκέ, που είναι η στη συγγήτριά μα, δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα αλλά μου είπε ότι για την τροπολογία 15 έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Επομένω δεν χρειάζεται πια χωριστή ψηφοφορία. Μα θέλετε σα διαβάζω το κείμενο το οποίο συμπεφωνήθη στα αγγλικά. Λέει, ενώ μια άνηση κατανομή σπάνιων πόρων μπορεί να εμποδίσει την καινοτομία, θεωρεί ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρώτες ύλες θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις κυρίες πρόκλησεις για να υπάρχει ισοδίκαια πρόσβαση στους πόρους αυτού. αυτούς. Αυτό είναι το κείμενο το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ψήφι πέρα αυτής της τροπολογίας, όπως έχει τροποποιηθεί, κατά, αποχές, δεκτή. 16. Ψήφι υπέρ της 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Κύριε Μπιτικόφερ, παρακαλώ. <clears throat> Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Μπιτικόφερ. Μικρόφωνο, παρακαλούμε. Για την 103 ε, εξέπεσε, είπατε, αλλά δεν κατάλαβα γιατί αυτή η τροπολογία. Επειδή καλύπτεται από την 2 της ΙΜΚΟ. ΙΜΚΟ 2. Στην ε, παράγραφο 22α νέα αναφέρεται ότι αν γίνει δεκτή η ΙΜΚΟ 2 τότε εκπίπτει 103. Εντάξει λέει ο κ. Μπουτικόφρα. Ε. Συνολική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Υπάρχει ένας ε, παραπάνω από τους βουλευτέ του ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίες. Σαφές το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον κύριο Βίνκλερ. πρόγραμμα Κοσλοντούι με την συγκεκριμένη την κυρία Χάρμς. Υπάρχει ο κατάλογος ψηφοφορίας, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα το κάνουμε στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Ξεκινάμε λοιπόν. 5. Πέντε της εισηγήτριας. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 32. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 εκπίπτει. Όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Η 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 31. Εκπίπτει. Εκπίπτει αν εγκριθεί η 5. 31, όχι, την ψηφίσουμε, υπέρ. Συγγνώμη, ήταν σωστό αυτό που σας είπα στην αρχή. Εκπίπτει γιατί είναι κρίθη 14. 30, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6, 6 έχει αντικατασταθεί από μια προφορική τροπολογία της ε, εισηγήτριας ψήφι υπέρ της προφορικής τροπολογίας κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 με χωριστή ψηφοφορία που από Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα της 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Σας το ξαναλέω. Πέρας. Όχι. Εντάξει. Πάλι. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Πάλι να δοκιμάσουμε. 16 τμήμα 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 37. Εκπίπτει, εκπίπτει. Πάω πολύ γρήγορα. Και τώρα πηγαίνουμε στην 38. Πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Θα το έλεγξω Πέρας. Εκ... Ε, απορρίπτεται. 17. 17 κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 και 18 ταυτίζονται ψηφί <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτές 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 Εκπίπτει, εκπίπτει αν έχει εγκριθεί η 6. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Δεν έχει εγκριθεί 6. Ψήφι υπέρ. 42. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Χωρίς την ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 44 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τώρα έχετε το δύσκολο. 8. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 8. Ψήφι υπέρ 8. Κατά αποχές δεκτή. Εκπίπτει η ανακατά συνέπεια 9 ψήφι υπέρ. Ψήφι υπέρ της 9 κατά αποχές δεκτή. 1 της εισηγήτριας ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτωτη. 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 <coughs> Ψήφι Κατά. Απόχες. Δεκτή. <coughs> Τρία ψήφι <coughs> Κατά. Απόχες. Δεκτή. Δεκατέσσερα ψήφι υπέρ σε δύο τμήματα. Έχουν εκπέσει οι προηγούμενε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Πω, πω, ξέχασα τη συμβαστική ένα λέει. Μεα κούλπα. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Το είχα ξεχάσει αυτό το πράγμα. 14. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. το τμήμα εκπίπτει. Εκπίπτει, γιατί είχε απορριφθεί το πρώτο τμήμα. Μάλιστα, ωραία. Πέντε περιβάλλον. <clears throat> Εκπίπτει. Όχι. Όχι, την πέντε την ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Συμβαστική 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Όχι, όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, ξέχασα την τροπολογία 25. 25 τροπολογία ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές απολύτωται. έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος είναι 28 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 <clears throat> ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 12. Περιβάλλον υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 προϋπολογισμόν υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 προϋπολογισμόν υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 προϋπολογισμόν κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Ανοιχτή, ανοιχτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Τέλος, το νομοθετικό ψήφισμα. Πάλι ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα. Εντάξει, πάει και αυτό. Ενεκρίθη. Ε, συγχαρητήρια στην κυρία Χάμς. Ήταν δύσκολα όλα αυτά. Αλλά πέρασε η έκθεσή σας, αλλά ήταν δύσκολα όλα αυτά και σας συγχαίρω. Κύριε Χάνς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που δίνετε και πάλι το λόγο κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Ίσως είδατε ότι καταψήφισα την έκθεσή μου και η ομάδα μου το ίδιο εδώ. Το έκανα χωρίς να είναι και η πρόθεσή μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η όλη συζήτηση, αλλά υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν έχουν επιληθεί τα θέματα των αποβλήτων από το Κοσλοντούι και είναι σαφές ότι στην ε, Βουλγαρία δεν υπάρχει καμία χρηματοδοτική πρόβλεψη για την εναπόθεση των αποβλήτων. Τα απόβλητα θα εξαχθούν από τη Βουλγαρία στη Ρωσία. Αυτό είναι μονόδρομος πια αυτή η διαδικασία και για μένα η συζήτηση αυτή ήταν πολύ σημαντική σε σχέση με την ε, προετοιμασία της οδηγίας για την τελική κατάργηση πυρηνικών σταθμών της Κομισιόν και το δεύτερο τμήμα της συζήτησης αφορούσε το θέμα του γιατί δίνουμε τόσα πολλά εκατομμύρια στη Βουλγαρία νοπό χρήμα εάν δεν εξυπηρετούν πραγματικά το στόχο της κατάργησης των πυρηνικών σταθμών στο Κοσλοντούι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν για τις ανανεώσιμες ενέργειες και την, ε, το εξυγχρονισμό των δικτύων διανομής ενέργειας. Αυτό θέλησα να περάσω σε αυτή την Επιτροπή, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Επιτροπής μας δεν δέχτηκε κάτι τέτοιο. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να επανέλθουμε στην Ολομέλη και να ξαψηφίσουμε, αλλά θα ήθελα να γίνει σαφές σε όλες τις πολιτικές ομάδες κατά πόσο υπήρξε και μεγαλύτερη υποστήριξη στην αρχική μου αίτηση και από άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέω πρόεδρος, για την διευκρίνησή σας. Τώρα ξέρουμε όλοι γιατί ψηφίσατε έτσι. Τελειώσανε λοιπόν οι ψηφοφορίες και μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σημείο 9. Ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης. Ο κύριος Ρέμεκ είναι ο αρμόδιος. Ναι, παρόν. Είσαστε εκεί. Κύριε Ρέμεκ, έχετε το λόγο. Θα χαρούμε πάρα πολύ εάν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση να μην ενοχλούν τον κύριο Ρέμεκ και να αποχωρήσουν ηρέμως και ησύχω. Όποιο δεν ενδιαφέρεται λοιπόν για τη δορυφορική πλοήγηση να αποχωρήσει ταχαίω και ηρέμος. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να συνεχίσετε τα πηγαδάκια σα έξω και να συζητήσετε ό,τι θέλετε και να μας αφήσετε και εμάς να συζητήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, στο σημείο 9 αρχίζει η συζήτηση. Κύριε Ρέμεκ, έχετε το λόγο. Έχετε το έγγραφο εργασία στου φακέλου σα, οπότε εγώ δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μονάχα μερικέ παρατηρήσει. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι η μόνη η οποία θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα δορυφορική πλοήγηση. Οι πληροφορίε δείχνουν ότι υπάρχουν και άλλε σημαντικέ χώρε σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίε είναι ανταγωνιστικέ σε, εμά, σε εμά, με εμά, με την Ευρώπη, που αυξάνουν τι προσπάθειε στον τομέα αυτό, όχι μονάχα οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία, αλλά και χώρε όπω η Κίνα και η Ινδία. Έχουμε τον ανίβα πρώτων θυρών, λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατεπηγόντως το θέμα αυτό. Ο στόχο αυτή τη έκθεση είναι να εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων και πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και να προχωρήσουμε επιτυχώ στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, το οποίο είναι δάπανο φυσικά και πολύπλοκο. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε συσσωρεύσει καθυστερήσει, έχουμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να βρούμε του μηχανισμού και συστήματα χρηματοδότηση για το, τη δορυφορική πλοήγηση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και δομέ διαχείριση και εξάλλου δεν είμαστε απόλυτα ανεξάρτητοι σε ό,τι αφορά την εκτόξευση και την διαχείριση των δορυφόρων. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστος και σε τελική ανάλυση οι ανταγωνιστές μας βελτιώνουν τις τεχνολογίες τους και προχωρούμε μεγαλύτερη ταχύτητα με την Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα κάποια βεβαιότητα η οποία πλανάται σε πολιτικό επίπεδο, διότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αμφιβολίες αν θα υπάρξει υποστήριξη προγραμμάτων όπως ο Γαλιλαίος. Ο δικός μου στόχος ως ενδιαφερομένου και εμπλεκομένου σε αυτό το σχέδιο είναι όλες οι ιδέες αυτού του ευραίου φάσματος πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο να αντανακλώνται στην εκθέσή μου. Επομένως θα προσπαθήσω να συλλέξω όλες τις παρατηρήσεις σα, όλες τις συστάσεις και τις ιδέες σα στην εκθέσή μου για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα αποδεκτό για όλους. Θα με ενδιέφερε να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε για να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου ενός ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης με δορυφόρο που να δίνει προσθέμενη αξία και να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρωτοπορία της τεχνολογίας ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά μας και να υποστηρίξει την οικονομία και την απασχόληση και να συμβάλλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα και μια υποδομή που να είναι στερεά αυτή η υποδομή και εύρωστη και να επιτρέψει να υπάρχει μια προσφορά υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Δεν αφορά μονάχα ένα συγκεκριμένο χώρο δραστηριοτήτων, αφορά όλε τι δραστηριότητε της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι η Ευρώπη χρειάζεται αυτό το σύστημα και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεπεράσουμε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο πρόεδρο. Κυρία Χόλτσερ, έχετε, λάβει το, ζητήσει το λόγο. Κυρία Χόλτσερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος ε, τον κύριο Ρεμέκη για αυτό το έγγραφο εργασίας. Είναι σαφέστατο και μας βοηθάει με τον τρόπο που το παρουσιάζει γιατί θέτει τα σωστά ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που αναφέρει στο εγγραφό του. Τα συζητήσαμε το πρωί με τον Επίτροπο κάποια από αυτά, αλλά δεν πήραμε απαντήσεις. Ελπίζω ε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας ε, να τα καταφέρουμε καλύτερα, να βρούμε κάποιες απαντήσεις. Αναρωτιέμαι αν ε, θα έπρεπε να αναλύσουμε εντελεχώς ακριβώς ποια θα είναι τα, ποιοι θα είναι οι καρποί του Γαλιλαίου. Μέσα στο έγγραφο εργασίας ε, καταδεικνύεται ότι δεν υπάρχει πλέον εμπορικός ρόλος για τον Γαλιλαίο. Έχει σημειωθεί τόση μεγάλη καθυστέρηση που τώρα είναι σε ανταγωνισμό με διάφορα συστήματα, το κινέζικο, το ιαπωνικό, από τεχνολογικής δε δεν είναι στην αιχμή της τεχνολογίας όπως έλεγα. Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής υποδομής, δηλαδή εντάξει θα έχουμε μια ευρωπαϊκή δορυφορική ικανότητα. Αλλά αν έτσι το δούμε ως πρόγραμμα υποδομής, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε αν αξίζει εφόσον ε, έχουμε περιορισμένους δημοσιονομικούς πόρους. Μα τι καρπούς θα αποφέρει, τι περιμένουμε από αυτό σε σχέση με άλλα είδη υποδομών στα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένω να επενδύσουμε αντί για τον Καλλιλέο. Ε, κάποια πράγματα δεν ε, να αναφέρονται καν ε, στο έγγραφο. Ε, δηλαδή όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε το Γκαλιλαίο και υπέγραψε αυτή την συμφωνία ιδιωτικού δημόσιου τομέα, τόνισε ότι είναι... ότι δεν είναι στρατιωτικό σχέδιο Και ξαναλέω ότι τώρα πια από εμπορική πλευρά φαίνεται ότι έχει χάσει την αξία του τον Γαλιλαίο. Δεν πρέπει να το αναφέρουμε αυτό μέσα στην έκθεση. Ε, υπάρχουν και γκρίζε ζώνε εξάλλου κατά τη χρήση του. Παραδείγματο χάρη ασφάλεια για τι ε, επιχειρήσει ε, διατήρηση ειρήνη. Δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ αυτά και όλο το αποφεύγουμε το θέμα. Έχει, ε, έχουμε απολέσει τον αρχικό στόχο του Γκαλιλαίου πλέον, αυτό εννοώ και διάφορε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον Γαλλίο για άλλε σκοπιμότητε πλέον. Επίση αναρωτιέμαι για την ασφάλεια ε, του προγράμματος από δύο πλευρές. Η τεχνική, ε, η τεχνολογική ασφάλεια λόγω φυσικών φαινομένων ε, και όλοι το είδαμε πριν από λίγους εβδομάδες ότι πάτε μας ξαφνιάζει η φύση ε, για τη μείωση της ε, ακτινοβολίας, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να καταρρύψει τους δορυφόρους, ε, να τους βγάλει off. Υπάρχει φεδρικό σχέδιο, εν τη περιπτώσει έχουν εξετάσει αυτόν τον κίνδυνο καν. Ε, γιατί αν αρχίσουμε να εξαρτώμαστε από το σύστημα πρέπει να κατανοήσουμε ε, ποιοι είναι οι φυσικοί περιορισμοί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουμε. Τώρα ε, η πολιτική σκοπιά του ζητήματος δεν απάντησε ο Επίτροπος το πρωί αλλά στην ακρόασή του όταν το ρωτήσαμε για το ρόλο της Κίνας που υποτίθεται ότι συνεργάζεται μαζί μας με την ιδιότητα του εταίρου για τον Γαλιλαίο αλλά τελικά αρνείται να παραχωρήσει τη χρήση του δικού τους κομματιού του ε, ραδιοφάσματος ε, στα πλαίσια του προγράμματος Γαλιλαίο και αυτό σαφέστατα ε, αναδεικνύει το λένε και περισσότερο σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. Θα ήθελα να ξέρω αν έχουν σημειωθεί εξελίξεις για αυτό το θέμα από την ακρόαση του Ιανουαρίου μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα. Τι δράση αναλαμβάνετε, πώς θα Ε, το μεθοδεύσει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, ε, το θέμα της εμπλοκής της Κίνας δηλαδή στο όλο πρόγραμμα. Τέλος, ε, είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος, κοινοβουλευτικός έλεγχος για αυτό το θέμα. Έχουμε την ε, συμβαστική συμφωνία ε, βάσει της οποίας ε, ένας βουλευτής μπορεί να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή σήμερα προσφέρει να χρησιμοποιεί περισσότερο την ε, διαδικασία αυτή. Οπότε ζητώ να έχουμε ε, τα έγγραφα αρκετά πριν από τις συνεδριάσεις ε, γιατί μέχρι στιγμής τι γίνεται, τα παρουσιάζουν όταν γίνεται το Συμβούλιο, οπότε δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για ανάλυση των εγγράφων και προετοιμασία από πλευράς του Κοινοβουλίου. Οπότε εφόσον επιδιώκουμε ε, αυξημένο δημόσιο έλεγχο, πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Ε, ξαναλέω ότι ο συγητή μα βοηθά με την ανάλυση που κάνει μέσα στο έγγραφό του και με ικανοποιεί πάρα πολύ η παρουσίαση του ζητήματο ε, και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμεί αποτελεσματικότερα στην έκθεση. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Γκλάντε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο κύριος Ρέμεκ έχει θέσει πολύ σημαντικά ερωτήματα μέσω από την έκθεσή του και η κυρία Χόλτα έχει θίξει και αυτά τα θέματα, οπότε μπορώ να είμαι σύντομο. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό τη χρηματοδότηση. Δεν είναι γενικά πρόβλημα μόνο για τον Καλλιλέο, αλλά και για το ΕΜΕΣ, που πρέπει να υπάρξει κάποια λύση. Πριν από μία εβδομάδα είχε συζητηθεί το τι μπορεί να κάνει κανεί για το προπολογισμό αυτού του εγχειρήματο. Θα υπάρξουν 14 δορυφόροι που θα εκτοξευθούν που είναι η πρώτη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει κάποιο είδος συνεργασίας μεταξύ του Γαλιλαίου και του GPS μπορεί κανείς να έχει πλοήγηση αυτοκινήτων με δορυφόρο από το Αμβούρο να πάει στο Χόλμ χάρη, αλλά δεν έχουμε τις άλλες υπηρεσίες παραγωγός χάρη, τις υπηρεσίες διάσωσης πλοίων στον από πλοία στον ωκεανό. Έχουμε μια ακρίβεια εντοπισμού της τάξης των 300 μέτρων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι επαρκή αυτή τη στιγμή. Και επίση έχουμε συζητήσει και με την Κίνα. Προσπαθήσαμε πριν από μερικά χρόνια να έχουμε καλύτερη συνεργασία με την ε, Κίνα και ξέρουμε τελικά ότι οι συνάδελφοι από την Κίνα θέλουν να πάρουν τεχνολογία από εμά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας. Υπάρχουν κάποια επίσης εξαρτήματα τα οποία θα παίρνουν από την Κίνα τα οποία δεν είναι πια ε, σύγχρονα, έχουν ε, γίνει πια πεπαλιωμένα. Οπότε δεν ε, μπορούμε να επωφεληθούμε και επίσης υπάρχει το πρόβλημα της παράλληλης χρήσης των, του, ίδιου, του ίδιου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από την Κίνα, το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Επομένως όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο Επίτροπος Ταγιάννη ήταν θετικά, αλλά θα ήθελα να έχω και πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Ξέρω φυσικά ότι δεν μπορούν όλα αυτά να δοθούν σε ανοιχτή συνεδρίαση και στη δημοσιότητα πλήρως, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πιο μικρό σώμα το οποίο μπορεί να πάρει σε εμπιστευτικό επίπεδο περισσότερες λεπτομεριακές πληροφορίες, ώστε να υπάρξει μια δυνατότητα να έχουν η αρμόδιοι δυνατότητα να γνωρίζουν τι γίνεται και να υπάρξει η απαραίτητη συνένεση των πολιτικών ομάδων για το εγχείρημα αυτό, κύριο Πρεζίνα. εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί κυρίως ο, οι σκιώδεις εισηγητές βοήθησαν πάρα πολύ να επιληθούν πολλά ζητήματα που ήταν εκκρεμή. Εγώ συμμερίζομαι αυτή την άποψη λοιπόν που αναφέρθηκε προηγουμένως σε σχέση με τις αμφιβολίες που ακόμα πλανώνται. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία για τα οποία θα ήταν χρήσιμο να είμαστε επίμονοι πριν προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτού του συστήματος. Πρώτα απ' όλα <clears throat> τίθεται το θέμα των τεχνικών και τεχνολογικών γνώσεων. Απαιτείται ένα σύνολο από γνώση σε αυτό το σχέδιο και εξάλλου δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η ανεξαρτησία των συστημάτων αυτών που αναπτύσσονται εκτός Ευρώπης. Και αυτά τα συστήματα δεν είναι 100% ανεξάρτητα. Τα συστήματα αυτά <clears throat> χρησιμοποιούν <clears throat> και στοιχεία τα οποία δεν είναι μονάχα πολιτικού χαρακτήρα αλλά και στρατιωτικά. Επομένως εμείς περιμένουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περισσότερα στοιχεία ιδίως από την Κομισιόν και πιστεύω ότι η Κομισιόν είναι αυτή η οποία θα πρέπει να προωθήσει περισσότερο τη συζήτηση αυτή. Είναι απαραίτητο λοιπόν, είναι απόλυτα υποχρεωτικό αυτό το σύστημα πλοήγησης μέσω δορυφόρων να κατασκευαστεί και να είναι εποφελής η Χριστού. Και νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Κύριε Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τον ε, κύριο Ρίμεκ, γιατί μέχρι στιγμή δεν είχα αφιερώσει χρόνο για να διαβάσω το έγγραφο εργασία του. Δηλαδή θα τον ευχαριστήσω, ναι, μένα, αλλά δεν το έχω διαβάσει ακόμη. Εάν έπρεπε να πάρουμε απόφαση σήμερα για το πρόγραμμα, Πιστεύω ότι δεν θα δίναμε συγκατάθεση. Έχουμε καθυστερήσει και πρόκειται για ε, ε πολλά χρήματα. Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι αρχίζουμε ε, από το μηδέν. Ότι έχει δρομολογηθεί το πρόγραμμα και δεν μπορούμε τώρα να υπαναχωρήσουμε. Ε, ας αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τότε αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Ε, θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση. Να πούμε ναι, είναι, λένε κάποιοι ότι είναι περιττό το σύστημα. Α δούμε για ποιες εφαρμογέ μπορούμε να διαφοροποιηθούμε από τι υπηρεσίε που προσφέρουν ανταγωνιστικά συστήματα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερον, από πλευρά διαδικασία, ε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα είναι το πρώτο βιομηχανικό πρόγραμμα που ε, θα διαχειρίζεται ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή θα το εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ από αυτή την οπτική γωνία βλέπω το σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένες φορές έχουμε την εντύπωση ότι, είναι, ότι υποστηρίζει την ενωσιακή δράση σε πολλούς ε, τομείς εναντίον όλων, οπότε τι θέλω να πω. Να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούμε να συνδιαχειριστούμε το σύστημα και έτσι θα ανοίξουμε τον δρόμο και για άλλα συστήματα. Οπότε από πλευρά διαδικασία ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα το ε, κλείσουμε ε, λαφρέα την καρδία όπω έκανε το έλκτο σύστημα. Να δείξουμε στην Επιτροπή ότι μπορούμε να έχουμε την κοινή διαχείριση γιατί αλλιώς ε, θα φανούμε ανόητοι με την ε, μέχρι του δεστάση μας. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο σημαντικές παρατηρήσεις όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Ταυσνόφσκι. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά τα οποία ακούστηκαν ε, για τον κύριο Ρέμεκ. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα τόσο υψηλού κόστους πρόγραμμα, καλό θα είναι να πετύχει, να θεωρηθεί επιτυχές. Έγιναν κάποια λάθη στην αρχή του προγράμματος, όταν είχε υποθεί ότι το σύστημα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ανταγωνιστικό και θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το αμερικανικό GPS. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα οποία σας είπα. Νομίζω ότι έχει σημασία πάντως για μας να μην θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα επιπλέον σύστημα δορυφορικής πλοήγησης να θεωρήσουμε ότι ε, το σύστημα αυτό μπορεί να βοηθήσει και την έρευνα Για να το πετύχουμε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά όλες τις πληροφορίες τις οποίες θα μας δώσει το δορυφορικό αυτό σύστημα. Προφανώς και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αυτό και για λόγους ασφαλείας, άμυνας. Ξέρουμε ότι σε πάρα πολλούς τομείς έχουμε ελληματικές μορφές ενημέρωσης και δεν αναφέρομαι μόνο σε στρατιωτικά θέματα. Και για πολιτικά προγράμματα το πρόγραμμα αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αίσθησή μου είναι ότι το σχέδιο αυτό θα επηρεάσει θετικά πολλές πλευρές της ε, ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε το πρόγραμμα Γαλιλαίο σαν μια ευρωπαϊκή υποδομή πλέον, όχι ένα ανταγωνιστικό επιπλέον εμπορικό σύστημα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εγώ στην αρχή ε, είχα κάνει λάθος όπως και όλοι οι άλλοι θεωρώντας ότι είναι ανταγωνιστικό με άλλα τέτοια συστήματα αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Κύριε euh, Είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι μια αποτυχία του ιδιωτικού τομέα τον Galileo Διακόπτει ο κύριος Σόδη. Αμικρόφωνος είμαι, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι μια, συνιστά μια αποτυχία του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με το business plan που είχαμε. Τα έσοδα σε καμία περίπτωση δεν θα καλύψουν κάποιες ε, ιδιαίτερα ψηλέ παρακινδυνευμένες επενδύσεις. Πέφτει λοιπόν στον δημόσιο τομέα τη στιγμή που αντιμετωπίζει προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Επίτροπος βέβαια μας διαβεβαίωσε για την πολιτική του απόφαση και θα υπάρξει και μια έκθεση πρωτοβουλίας από πλευράς Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβεβαιώσει τους πολίτες και το Κοινοβούλιο, γιατί αν υπάρξει μια επιπλέον αποτυχία λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για τεχνολογικούς λόγους, διότι οι συχνότητες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτό θα είναι ένα σκληρό χτύπημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έτσι και αλλιώ τα βρίσκει δύσκολα. Υπάρχει λοιπόν θέμα πολιτικό. Το θέμα εδώ ξεπερνά τα επιστημονικά ή τεχνικά προβλήματα, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σαφής σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό που είναι κρίσιμο για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει εις πέρας μείζωνα θέματα. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μια μικρή παρατήρηση. Είπατε πολύ σωστά ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό σχέδιο. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα συμβεί αν αυτό δεν λειτουργήσει, θα δείξει ίσως κάποια πράγματα, θα έχει κάποιες επιπτώσεις για το κατά πόσο είμαστε σε θέση να επομιστούμε τέτοιου είδους προγράμματα. Δεν αφορά μονάχα το τωρινό αυτό πρόγραμμα. Επίσης, η πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί ξεκινώντας από το μηδέν. Το ερώτημα είναι παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό θέλω να θέσω αυτό το ερώτημα με την Κομισιόν. Μήπως θα πρέπει να έχουμε κάποιους νέους δορυφόρους και να συμπληρώσουμε το σχέδιο. Είναι ζήτημα κόστους. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι δύσκολα, η μια ανάλυση κόστους ωφέλειας, αλλά θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια σαφή πληροφόρηση από την Κομισιόν. τι γίνεται λοιπόν με τους πυράβλους φορείς. Τι είδους ε, πύραυλοι φορείς χρησιμοποιήθηκαν, επελέγησαν και, για, και πώς συνδέεται το κόστος με αυτά για την ε, τελική ανάλυση και για την χρήση του συστήματος. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο. Λοιπόν, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε αν θα μπορούμε να έχουμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε και πάλι για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα προηγουμένως να έχω και την άποψη της Κομισιόν και η κυρία Νίπλερ ίσως να λάβει το λόγο πριν από την Κομισιόν. Η Αγγέλικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που θέλω να πω στη συζήτηση τόσο καθυστερημένα. Αλλά αυτό το προκάλεσε και η δική σας παρέμβαση με έκανε να λάβω το λόγο γιατί αυτό το οποίο λέτε το βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγάλη σημασία να έχουμε ένα σαφές μήνυμα το οποίο θα στείλουμε όχι για το Γαλιλαίο συγκεκριμένα ή για κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα, αλλά αν εμείς στην Ευρώπη δεν μπορούμε να έχουμε αυτόνομη υποδομή για την πλοήγηση. Αυτό ίσως δεν μας δίνει πολλές δυνατότητες να μας παίρνουν στα σοβαρά και σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, ο Γαλιλαίος είναι έκφραση της θέλησης Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει το δικό της σύστημα πλοήγησης, όπως έχουν οι Αμερικάνοι, όπως οι Κινέζοι θέλουν να έχουν πολύ σύντομα, όπως θα κάνουν και οι Ρώσοι. Επομένως, αν εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα, αυτό σημαίνει και απώλεια διεθνούς βάρους για την Ευρώπη. Επομένως πρέπει εμείς να κάνουμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και να αποκτήσουμε αυτή την υποδομή. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι το μήνυμα το οποίο θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ερώτημα το οποίο θέσατε κύριε Πρόεδρε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τις λειτουργικές λεπτομέρειες τους πυράβλους φορείς και είναι χρήσιμο για τους άλλους συναδέλφους να εξασφαλίσουμε την υποστήριξή τους και γι' αυτό θα είναι απαραίτητο να έχουν τις πληροφορίες ώστε να δώσουν και αυτοί το ναι. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θέλει να λάβει το λόγο από εσά. <clears throat> Κάπως ε, αυθόρμητα το αποφασίσαμε με ο κύριος Σμιτ, το άτομο το οποίο δεν ε, έπρεπε να λάβει το λόγο, έχασε την κάρτα του και δεν μπορούσε να μπει στο κοινοβούλιο. Είχε πρόβλημα να μπει. Ορίστε, δεν μπορεί να έρθει ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν εδώ στη συζήτησή μα γιατί δεν είχε την κάρτα του. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, σα ακούω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω το ερώτημά σα λέγοντα το εξή, λέγομαι Μπέρνα Σνίτκερ, είμαι στα πλαίσια του συστηματο αυτού Γαλλίου, με γνωρίζουν ορισμένοι από εσά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να, λάβετε το, να λάβω το λόγο εδώ. Υπήρξαν ορισμένες παρεμβάσεις ήδη για ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουν και νομικό χαρακτήρα εν μέρη, αλλά θα προκαθορίσουν και το μέλλον του Γαλιλαίου αν θα πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα ναι ή όχι. Αυτό το ερώτημα όμως θα έπρεπε να έχει τεθεί πριν από 2,5 χρόνια όταν ζητήθηκε να υπάρξει η χρηματοδότηση για την αρχική βάση του σχεδίου, δηλαδή να δημιουργηθεί το βασικό πλαίσιο των δορυφόρων. Αυτό θα έπρεπε ίσως να τεθεί το ερώτημα τότε. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε με το σχέδιο αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε δώσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μετά να πούμε όταν οι δορυφόροι εκτοξευτούν να τους ε, αλλάξουμε και να κάνουμε ένα νέο σύστημα και για κάτι τέτοιο δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Και οι πολίτες και η βιομηχανία περιμένουν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ότι εμείς στην Ευρώπη έχουμε την πολιτική θέληση να υποστηρίξουμε και να χρηματοδοτήσουμε μακροχρόνια ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτό σημαίνει και κατά τη διάρκεια των επομένων επτά ετών δημοσιονομικών προοπτικών αλλά και επέκεινα. Θα πρέπει λοιπόν η βιομηχανία να ξέρει ότι υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτό το σχέδιο. Επανέρχομαι τώρα στην έκθεση του κυρίου Ρέμεκ και στην, στο έγγραφο συζήτησης του εισηγητή. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση πρώτα. Μπορούμε να λάβουμε συγκεκριμένες θέσεις για το έγγραφο αυτό αλλά κάποιο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί στην προβληματική είναι το θέμα της οικονομικής χρησιμότητας του Γαλιλαίου και εδώ έρχομαι στις παρατηρήσεις της κυρίας Χολ. Πράγματι σήμερα θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα σε σχέση με άλλα σχέδια ή με άλλα εγχειρήματα τι θα προσφέρει το Γαλιλαίο, τι θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσουμε χρηματοδότηση στο Γαλιλαίο ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα υποδομής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το έχει αντιμετωπίσει ήδη η Κομισιόν από τη δική της πλευρά. Ο κ. Σταγιάννη ανέφερε σήμερα το πρωί ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό της ε, οικονομικής ωφέλειας από το Γαλιλαίο σε σχέση με το κόστος να το συζητήσει. Έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε συλλέξει πληροφορίες Απλώς θα ήθελα να πω εν μεγάλη συντομία ότι κατά τη δική μας άποψη το Γαλιλαίο δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μονάχα σαν ένα πρόβλημα χρηματοδότησης, αλλά σαν ένα ατού το οποίο μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική της ανάπτυξη και επομένως δεν είναι χρήματα που τα από το παράθυρο, δεν είναι υποδομές που δεν εξυπηρετούν κανένα ρόλο είναι αντίθετα μια υποδομή η οποία θα προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θέσεις απασχόλησης, ακόμα και σε άειλες, άειλης μορφής πρόοδο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα τονίσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς από την πλευρά της Κομισιόν με τις δικές μας ανακοινώσεις και ο κύριος Ρέμεκα ελπίζω με τη δική του έκθεση θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Γαλιλαίο έχει μεγάλη ωφέλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Για την οικονομική πλευρά Επομένως είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλες διαστάσεις που είναι σημαντικές, η μη οικονομική διάσταση, η δυνατότητα της Ευρώπης να καταδείξει ότι μπορεί πράγματι να στήσει ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα και εκεί η κυρία Χολ έχει αναφερθεί, είπε ότι δεν πρόκειται για, για μια τεχνολογία εχμής στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γαλιλαίου, ιδίως ό,τι αφορά τα ατομικά ορολόγια, αλλά αυτό το οποίο είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα αυτού του σχεδίου. Πολύ λίγοι φορείς, πολύ εσοντότητες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αυτή την ικανότητα και η Ευρώπη θα πρέπει να καταδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να δαμάσει αυτή την πολυπλοκότητα και δεν αναφέρομαι τώρα σε άλλα στρατηγικά θέματα αν θέλουμε οι τράπεζες, οι επικοινωνίες της Ευρώπης να υπόκεινται σε μία, να εξαρτώνται από μία υποδομή την οποία δεν ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο υποβόσκει σε όλη αυτή την προβληματική <clears throat> και πιστεύω ότι και αυτό το θέμα θα μπορούσε να το διεξέλθει ο εισηγητής σας, ο κύριος Ρέμεκ. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θίγει ο εισηγητής ο κύριος Ρέμεκ και αυτά μπορώ να τα αντιμετωπίσω εάν έχω τον απαραίτητο χρόνο. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Πρωτού ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Ρέμεκ, θέλω να υπενθυμίσω το εξή. Υπάρχουν χώροι για να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα όμως να έχουμε απέναντί μας ένα εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος είναι εμπειρογνώμων για τα θέματα αυτά. Και αυτό να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην μιλάμε στα περιθώρια του θέματος, αλλά να έχουμε μία μισή ώρα, μία ώρα για να, συζητήσουμε, να συζητήσουμε λεπτομεριακά για το θέμα αυτό και να πάρουμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μία συζήτηση με διερμηνία και με παρουσία όλων των συναδελφών. Να γίνει στην αρχή, στο τέλος μια συνεδρία, ώστε να είναι παρόντες όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μονάχα, αλλά σας λέω ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα η οποία πλανάτε, ενώ παράλληλα και εσείς τονίσατε ότι αυτό είναι ένα δυνητικά πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο. Ίσως λοιπόν πρέπει να καθορίσουμε και κάποιο ραντεβού τις επόμενες εβδομάδες, ώστε τα θέματα αυτά τα οποία υπάρχουν, συν τα πρόσθετα ερωτήματα τα οποία μπορούν να θίξουν οι συνάδελφοι, να απαντηθούν. Δεν χρειαζόμαστε επιτρόπου. Εδώ χρειαζόμαστε κάποιον στην Επιτροπή ο οποίο έχει γνώση των τεχνικών θεμάτων για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το σύνολο αυτών των ζητημάτων με ακρίβεια. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσεί ότι για την έγκριση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε επακριβώ περί τίνο πρόκειται. Η κυρία Χόλ λοιπόν και θα δώσουμε μετά το λόγο στον κύριο Ρέμεκ. Έχετε το λόγο κυρία Χόλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν και διαφοροποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιους τομείς, σε άλλους συμφωνούμε μαζί της. Το τομέα της ασφάλειας του συστήματος, σε σχέση με φυσικές καταστροφές ή το τι συμβαίνει με την Κίνα είναι κάτι το οποίο δεν απαντήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απουσία του υπεύθυνου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δύσκολο να πάρουμε απάντηση. Αν είναι όμως δυνατόν να μας ενημερώσετε ιδιαίτερα τι γίνεται με την Κίνα. Το θέμα είναι αν απελευθέρωσαν το φάσμα συχνοτήτων, ναι ή όχι. Ναι, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έφτασε, βρήκε την κάρτα του, αλλά δεν άκουσε τις ερωτήσεις δυστυχώς. Η είσοδος ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι λίγο δύσκολη για αυτούς που έχουν ξεχάσει την κάρτα τους, αλλά θα τα καταφέρω καλύτερα στο μέλλον. Για την Κίνα πριν να δώσω απάντηση να ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας. Θέλουμε να απαντηθούν οι ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν μπορεί η γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να συγκεντρώσει τις ερωτήσεις τις οποίες έχουν τα μέλη, έτσι ώστε να σας δώσουμε μια τεκμεριωμένη απάντηση η οποία θα έχει γίνει αντικείμενο προετοιμασίας για την κατάσταση στην Κίνα και για το φάσμα συχνοτήτων. Οι συχνότητες γενικότερα αφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν συστήματα είτε επίγεια είτε διαστημικά και απαιτείται μια συνεχής διαπραγμάτευση. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ληφθεί μια απόφαση, έχει τερματιστεί το σέμα γιατί τα περισσότερα συστήματα για διάφορους λόγους θέλουν να αλλάξουν και πρέπει να βρεθούν λύσεις και για, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγορών χωρίς να παρεμποδίζονται και να τυφλώνονται οι δυνατότητες των άλλων και θα πρέπει τα συστήματα να είναι λειτουργικά. Αυτή είναι η γενική διαδικασία θα έλεγα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ναι μεν από τη μία δεν πρέπει να υπάρξουν, να υπάρχουν παρεμβάσεις στο σύστημα, αλλά υπάρχει ένα θέμα με τις ε, κρατικές, κρατικά μηνύματα, αν τις κρατικές συχνότητες για λόγους εθνικούς ασφαλείας. Αυτά αποφασίζονται με διμερείς συμφωνίες, εκτός των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται να γίνονται στις στα Ηνωμένα Έθνη ή σε άλλες διεθνείς τηλεπικοινωνιακές οργανώσεις. Κάνουμε λοιπόν τέτοιες συζητήσεις με την Κίνα, τη Ρωσία, τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Ιαπωνία και την Ινδία. Με τις Ηνωμένε Πολιτείε κληρώθηκαν ε, επιτυχώς. Υπήρξαν συμφωνίες οι οποίες προστίθενται ε, επιμέρους τεχνικές συμφωνίες τη γενικότερη συμφωνία που έχουμε με τη ΣΥΠΑ και συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους. Η κατάσταση με την Κίνα παραμένει δύσκολη. Ξέρετε ότι έστειλε επιστολή ο πρόεδρος Μπαρόσο στον πρωθυπουργό της Κίνας έτσι ώστε να βρεθεί μια κάποια λύση. Θα υπάρξουν τεχνικές συναντήσεις πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά παραμένει το πρόβλημα περίπλοκο λόγω του ότι δεν καταφέραμε ακόμα να προχωρήσουμε στο παρελθόν και τα δύο συστήματα έχουν προχωρήσει σε επίπεδο προμηθειών και αν πρέπει να υπάρξουν ε, γενικά παραχωρήσεις από τη δική μας ή από την άλλη πλευρά, αυτό σημαίνει αλλαγές στις υποδομές και στους εξοπλισμούς, κάτι το οποίο θα κοστίσει ιδιαίτερα. Όλοι μπορούν να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις για να λυθούν τα προβλήματα, αλλά στην πρακτική αυτό είναι δύσκολο. Κάναμε κάποιες προτάσεις στους Κινέζους για το πώς θα βγούμε από το περίπλοκο αυτό ε, επίπεδο συνομιλιών. Απαιτείται να υπάρξουν λύσεις γρήγορα, γιατί εμείς βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια λειτουργίας του Γκαλιλαίου και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχουμε προχωρήσει ικανοποιητικά, τότε το θέμα μπορεί να προκαλέσει μια κάποια μορφή κλιμάκωσης το θέμα είναι ότι οι μηχανικοί, οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί θα πρέπει να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν να δουν τι αλλαγές θα πρέπει να υπάρξουν σε επίπεδο ηλεκτρονικών υποδομών. Και γι' αυτό ακριβώς έστειλε την επιστολή ο πρόεδρος Μπαρόσο, έτσι ώστε ε, να ενημερωθούν πολιτικά από την ηγεσία τους ε, οι αρμόδιοι σε επίπεδα τεχνικά. Η κατάσταση στην Κίνα είναι βέβαια περίπλοκη, γιατί υπεύθυνο για όλα αυτά είναι το κόμμα ή μάλλον είναι ο λαϊκός στρατός, το People's Liberation Army, ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Και είναι περιορισμένοι οι τρόποι επικοινωνίας που μπορεί να έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το PLA, με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάστηκε να έρθουμε απευθεία σε επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν ξέρω αν θέλετε απαντήσει σήμερα σε άλλες από τις ερωτήσεις σας θα πρέπει να μου τις θέσετε τώρα ξανά. Η Νίμπλα. Όχι είναι. Ο κύριος Ρέμεκ. Ίσως ε, να μην είναι δυνατόν να δοθούν ε, απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ένα τμήμα των ερωτήσεων μόνο έχει απαντηθεί. Ε, έχουν γίνει πάντως αρκετές προτάσεις όπως αυτή για την οργάνωση μιας συγκεκριμένης συνάντησης των μελών της Επιτροπής μας και μελών άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών που ενδιαφέρονται ή εμπλέκονται με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Ε, σαφώς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε μια τέτοια συνάντηση για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να σταθώ λίγο σε αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος Νίμπλα. Η επιχειρηματολογία της υπέρ του Γαλιλαίου μου φάνηκε ιδιαίτερα ελκυστική Παράλληλα με όλες τις άλλες συναντήσεις οι οποίες έχουν οργανωθεί, πήρα μέρος και σε μία συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Συστήματος GPS. Η συνάντηση αυτή έγινε off the record, δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά είχα θέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Εγώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής είχα ρωτήσει αν υπάρχει δυνατότητα για ένα πραγματικά διεθνές σφαιρικό πρόγραμμα πλοήγησης. Απάντησε ότι θεωρητικά θα μπορούσε να είναι εφικτό ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όταν ρώτησα ποια είναι τα εμπόδια σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, έτσι ώστε το GPS να είναι στη διάθεση ελεύθερα χωρών όπως και της Κίνας, απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να μοιραστούμε όλα τα επίπεδα πληροφοριών με όλους ανεξαρτήτως τους εταίρους Ρωσία, Κίνα κτλ. Δεν αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από το ύφο του, από τη διατύπωσή του κάτι τέτοιο νομίζω ότι ήταν ε, σαφές. Λοιπόν, στην Κίνα και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή προχωρούν στην διαμόρφωση τέτοιων τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερως επικαιροποιημένε. Υπάρχει επιθυμία επίσης από πλευράς και άλλων χωρών για να πάρουν μέρος στη διαμόρφωση αυτού του συστήματος και να καλύψουν και τις ανάγκες τους στον τομέα της ασφάλειας και αναφέρουμε εδώ ασφάλεια στρατιωτική. σχετικά με τις φυσικές καταστροφές. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο θα έπρεπε όλοι να είμαστε δεκτικοί και ανοιχτοί. Θα πρέπει όμως να υπάρξει και εδώ μια κοινή υποδομή, το κόστος της οποίας για την έναρξη λειτουργίας της θα υποστηριχθεί από πάρα πολλού. Το τούνελ του Μπρένερο σαν παράδειγμα κόστισε άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων. Προφανώς εγώ δεν είμαι κατά τον τούνελ, αλλά είναι ένα παράδειγμα αν θέλετε ανάμεσα σε άλλα υπερβολικού κόστους ε, περιφερειακών ε, προσπαθειών. Λοιπόν και εδώ χρειάζονται περισσότερα χρήματα από όσα είχαμε προβλέψει αρχικά για τη σωστή λειτουργία του Γκαλιλαίου. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς μένει να κάνουμε. Στην Τσεχική Δημοκρατία, σαν παράδειγμα, το πρόγραμμα Γκαλιλαίο θα κοστίσει πάρα πολύ και η Τσεχική Δημοκρατία ε, είναι διατεθειμένη να καλύψει το κόστος το οποίο της αντιστοιχεί. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι αξίζει τον κόπο να στείλουμε τα κατάλληλα μηνύματα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ανοιχτά. Συμφωνώ με όλους υποστηρίζουν την ιδέα εναρμονισμού του τρόπου με τον οποίο έχουμε να λύσουμε τα προβλήματα του, ε, του Γαλιλαίου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως έχουμε συμφωνήσει, οι πολιτικέ ομάδε έχουν την ευκαιρία στι επόμενε οι οποίες θα δοθούν στη γραμματεία και μετά η τρει μέρε να διατυπωσουν ερωτήσει, οι οποίε θα δοθουν στη γραμματεια και μετα η γραμματεια θα τι διαβιβάσει στην Κομισιόν. Και θα προσπαθήσουμε μετά το ταχύτερο δυνατό μέσα στη μέση διαταξή μα, να βρούμε μια χρονική στιγμή ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά παρακαλώ πάρα πολύ την Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να μα δώσει πραγματικά επακριβεί αποφάσεις, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα, έχει νόημα αυτή η περαιτέρω επαφή μόνο αν θα πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα του Κοινοβουλίου να σα υποστηρίξει, αλλά θέλουμε τις απαντήσεις. Ο κύριος Σοντή. Να ξεκαθαρίσω κάτι, να αποδέκτε την Επιτροπή, έτσι. Μας είπε ο εκπρόσωπός της ότι πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, ε, σαφέστατα ο, Επίτροπο Μπαρό έδειξε πολιτική βούληση και δυσκολευτήκαμε να βρούμε συμβαστικέ λύσει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χρηματοδότηση των πρώτων τριών ευδή. Άρα μα λένε τώρα ότι πρέπει να περιμένουμε την πολιτική βούληση. Δηλαδή, ε, αυτό που χρειάζεται τώρα σήμερα είναι να προχωρήσουμε και άρα η τεχνική πραγματογνωμοσύνη των μηχανικών κτλ. θα πρέπει να μα δείξουν ότι δεν ε, είναι άσκοπη η προσπάθεια. Για μα είναι σημαντικό ε, ο κίνδυνο, δηλαδή αν αποτύχει τελικά το πρόγραμμα, των παλάκων και τώρα είναι στο στρατόπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικής βούληση. είναι θέμα τεχνογνωσίας και εκτέλεσης από πλευρά των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει αυτό το σημείο, έχουμε στο σημείο 10. Είναι η γνωμοδότηση για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Και εδώ θέλω να ε, σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες εκπίπτει στις 4 ε, Μαΐου το μεσημέρι, σας το λέω εξ αρχής. Και δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λάγκεν, για να μας κάνει μια παρουσίαση για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έχει καθοριστεί η προθεσμία για τις τροπολογίες, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω ή δυνατόν να παραταθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αυτή η προθεσμία. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα που σας ζητώ να δώσουμε δυνατότητα στους συναδέλφους μέχρι τις 7 Μαΐου να παρουσιάσουν τροπολογίες. Θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο να έχουμε τη δυνατότητα οι τροπολογίες αυτές να μπουν στον μήλο της ε, μετάφρασης, γιατί στις 31 Μαΐου θα πρέπει να, αποφασίσουμε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Θα ήταν, <clears throat> πιστεύω, εφικτό να έχουμε τις τροπολογίες στις 31 Μαΐου και εγώ θα καταθέσω τροπολογίες και νομίζω είναι για όλους μας πολύ καλό να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ωραία. Προπα... ήταν αυτές οι παρατηρήσεις. Αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Κέλενεν είναι ο κύριος εισηγητής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και εδώ το θέμα που μας απασχολεί είναι οι εκπομπές διοξίδου του άνθρακος από τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Η πρόταση της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος που είναι η αρμόδια επί ουσίας, ακολουθεί μια κατεύθυνση παράλληλη με αυτή την οποία ανέφερα εγώ, ότι δηλαδή η νομοθεσία θα πρέπει να επεκταθεί και στην κατηγορία νη 1 των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Υπήρξε τώρα μια... Υπάρχει η πρόταση αυτή λοιπόν η οποία ακόμα είναι υπό την αιγίδα της διαδικασίας της συνθήκης της νίκαιας αλλά έχει αλλάξει η νομική βάση με τη συνθήκη της Λισαβόνας και η πρώτη μου πρόταση είναι, όχι μονάχα χρησιμοποιώντας το άρθρο 150 παράγραφος 1 που αφορά το περιβάλλον, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την πρόσθετη νομική βάση, το άρθρο 192 και το 114 για την εσωτερική αγορά, που είναι ένα νέο άρθρο. Τώρα το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε αυτή τη ρύθμιση με μια νομική βάση περιβάλλοντος ή εσωτερικής αγοράς. Και η Κομισιόν ανέφερε ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν θέμα εσωτερικής αγοράς. Στην αιτιολογική μου έκθεση και στην πρότασή μου υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία ίσως θα ήταν χρήσιμο να τα αναφέρουμε. Μείωση της ταχύτητος με ε, κόφτες, με συσκευές που περιορίζουν την ανώτατη ταχύτητα. Βέβαια δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο μόνο με περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων. Είδαμε τι έγινε στην περίπτωση της Κοπενχάγης, είδαμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την αύξηση της εναέριας κατηγορίας και είπαν και οι εμπειρογνώμονες ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξοικονόμηση που μπορεί να γίνει με την μείωση της τελικής ταχύτητας. Έχουμε επίσης το θέμα της εφαρμογής αυτού του αυτής της οδηγίας. Πώς θα ελέγχεται η, η παραμονή κάτω από τις οριακές τιμές. Είναι 135 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο το έτος 2020. Αυτό είναι ο μακροχρόνιος στόχος. 175 γραμμάρια ενώ θα είναι 120 για τα ελαφρά ιδιωτικά οχήματα. Και εμεί έχουμε, όπως ξέρετε, εγκρίνει αυτή την οδηγία για τα αυτοκίνητα, τα ελαφρά αυτοκίνητα. Είπαμε 120 μακροχρόνιος στόχος και 175 για τα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα, αλλά αυτή τη διαφορά θα προσπαθήσουμε στην πορεία του χρόνου να την μικρύνουμε και εδώ έχετε όλη η προβληματική της ε, βαθμίας εισαγωγής ώστε να φτάσουμε ως το 2018 σε ένα επίπεδο 150 γραμμαρίων. Η Κομισιόν έχει προτείνει 135 συνολικό στόχο, τελικό στόχο και αυτό σημαίνει μια περαιτέρω σημαντική μείωση των εκπομπών για τα μικρά επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει κάποια πραγματική αιτιολόγηση για να υπάρξουν τόσο αυστηροί κανόνες για τα μικρά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως για να υπάρξει τόσο μεγάλη πίεση να μειώσουν τις εκπομπές τους. Έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα μιας σταδιακής εισαγωγής πιο αυστηρών προδιαγραφών, αλλά δεν πρέπει εμείς να επιβαρύνουμε τόσο πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικά προβλήματα για αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό τόνισα ότι ο στόχος μας θα είναι να φτάσουμε το έτος 2025 σε 140 γραμμάρια και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητήσει κανείς, αλλά πιστεύω ότι μια παράταση για την επίτευξη του στόχου είναι απαραίτητο να δοθεί. Δεν θα έχουμε ούτως ή άλλως την οριστική απάντηση για αυτό το νομοθέτημα. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε επαρκή χρόνο στη βιομηχανία για να προσαρμοστεί. Επίσης, τα οχήματα τα οποία παράγονται σε διάφορα στάδια. Υπάρχει ένας αρχικός κατασκευαστής που φτιάνει το σασί μονάχα και τον κινητήρα και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν διαφορετικές υπερκατασκευές. Στην αρχή η Κομισιόν ήθελε να έχει την πλήρη ευθύνη ο αρχικός κατασκευαστής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεταπικιλία υπερκατασκευών. Θεωρεί τώρα ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία ε, κατάλληλη μέθοδος για να αντιμετωπιστεί το θέμα ευθύνης σε σχέση με τους, όλους τους κατασκευαστές που εμπλέκονται. Τώρα μέχρι πότε θα υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Η Κομισιόν είπε ότι αυτό θα γίνει μέχρι το 2011, αλλά εγώ ζήτησα μια μεγαλύτερη ε, χρονική διάρκεια. Για τα πρόστιμα, η Κομισιόν ακολούθησε το υπόδειγμα για τον, ε, των ιδιωτικών αυτοκινήτων και ζητά ένα πρόστιμο 125 για κάθε πρόσθετο γραμμάριο ανά χιλιόμετρο, ενώ ήταν μονάχα 90 το, το όριο, μάλλον το πρόστιμο για τα αυτοκίνητα για κάθε πρόσθετο γραμμάριο. Ξέρουμε ότι η Greenpeace θέλει πιο αυστηρές προδιαγραφές, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την Greenpeace να καθορίζει την βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, για, την, για τις πιστώσεις, προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν πάρα πολύ περιορισμένες προτάσεις από την Κομισιόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν περαιτέρω ελαφρύνσεις για τα οχήματα αυτά. Η Κομισιόν προτείνει για, τους, για τις μικρές επιχειρήσεις 20.000 το χρόνο ως όριο. Εμείς έχουμε προτείνει 25.000 πιστεύουμε ότι αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να γίνει για τα αυτοκίνητα που παράγονται σε μικρή σειρά με ένα ιδιαίτερο, με ένα ιδιαίτερο μηχανισμό. Αν μπορώ να πω κάτι ακόμα, λοιπόν, για την πρόταση της Επιτροπής ε, Μεταφορών, ε, συγγνώμη, Περιβάλλοντος, έχει προταθεί, έχουν προταθεί τα 150 γραμμάρια ως μακροχρόνιος στόχος αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2011 θα πρέπει να υποβληθεί μια συγκεκριμένη πρόταση. Θα έχουμε από το 2015 επίση, όπως λέει η πρόταση, μείωση ε, μέχρι τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει Όλη η, η επιβολή προστήμων να βασίζεται στα 95 ευρώ για κάθε πρόσθετο γραμμάριο και όχι 125 γραμμάρια όπως προτείνει η Κομισιόν. Και να υπάρξει λοιπόν η εφαρμογή όλων αυτών των ε, κανόνων αλλά με μεγαλύτερο χρόνο για να υπάρξει αυτή η προσαρμογή. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε και από τους συναδέλφους να υποβάλουν προτάσεις εναλλακτικέ και θα τις ζητήσουμε τον ε, Μάιο. Οι σκιώδεις ηγητές και πρώτος ο κύριος Περίλο. Αχ, excuse me. Don't see him. I've looked to the left. Περίλο. Η γνωμοδότηση του κυρίου Λάγκεν προκαλεί ορισμένες τροπολογίες με τις οποίες συμφωνώ και αναφέρομαι εδώ στις εξαιρέσεις τις οποίες προτείνει ο συνάδελφος. 95 ευρώ αναγραμμάριο δηλαδή εκπομπής. Δεν καταλαβαίνω βέβαια πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο αυτό το τμήμα των αυτοκινούμενων, αυτοκινούμενων οχημάτων. Αντίθετα με την προηγούμενη οδηγία, η οποία προέβλεπε ότι από το 2025 θα έχουμε μια αμέση εκπομπή 240 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο και όχι 135 όπως προτείνεται τώρα. Το 135 μου φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο ότι τα ελαφρά εμπορικά οχήματα τα οποία είναι χαμηλής απόδοσης ε, ε, σε εκπομπές είναι πάρα πολύ λίγα αλλά έχει υπάρξει η πρόοδος ιδιαίτερα για τους κινητήρες που κινούνται με πετρέλαιο και όχι με βενζίνη. Υπάρχουν επίσης και αεροδυναμικές βελτιώσεις αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του σχήματος που έχουν τα οχήματα αυτά τα οποία φυσικά ε, μεταφέρουν, ε, ε, πρέπει να έχουν μια κάποια χωρητικότητα μεταφοράς προϊόντων και ένα συγκεκριμένο ύψος, οπότε αεροδυναμικά έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ότι η ανανέωση των εμπορικών οχημάτων δεν είναι ιδιαίτερα δυναμική, δεν παρουσιάζει την ίδια δυναμική σε σχέση με τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. 10 χρόνια, στα 10 χρόνια αντικαθίστανται τα οχήματα αυτά και ο κύκλος παραγωγής τους είναι ε, πολύ πιο ε, μακρύς από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις λοιπόν οι οποίες ε, να συνεισφέρουν όσο περισσότερο γίνεται στην μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Επ' αυτού θεωρώ ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στον τομέα αυτό. Είναι αλήθεια ότι και η έρευνα έχει ανάγκη από κάποιο χρόνο για να βρει ορισμένε λύσεις, τις κατάλληλες λύσεις, οι οποίες ε, να συνδυάσουν τους κύκλους παραγωγούς και τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Δεν μπορούμε να προτείνουμε σήμερα περιορισμούς ε, μακράς περίοδου, αν δεν έχουμε συγκεκριμένες μελέτες και προβλέψεις οι οποίες θα καθορίζουν σαφέστερα τους στόχους τους οποίους έχουμε. Η κατάσταση είναι αποσταθεροποιητική για τη βιομηχανία και διαφωνώ και με την τροπολογία 16 του συναδέλφου Λάγκεν, του εισηγητή, που εισάγει από το 2018 μια ετήσια μείωση 5 γραμμαρίων κατ' για να φτάσουμε στο 2025 στα 135 ή 140 γραμμάρια. Νομίζω ότι η μείωση αυτή θα πρέπει σίγουρα να γίνει σταδιακά, αλλά δεν μπορεί τεχνικά να είναι εφικτός αυτός ο τρόπος ετήσιας μείωσης. Να θυμίσω ότι η παραγωγή ενός τέτοιου ελαφρού εμπορικού οχήματος ε, απαιτεί τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οπότε η ετήσια μείωση διοξιδίου του άνθρακα θα έλεγα δεν είναι εφικτή και δεν πρέπει να υποστηρίξουμε την τροπολογία 16. Ευχαριστώ κυρία Χόλα, το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν για την έκθεσή του. Ε, θα έλεγα ότι είμαι λίγο πιο ε, αισιόδοξη για την αυτοκίνητο βιομηχανία σε σχέση με τα ελαφρά οχήματα. Ε, πιο αισιόδοξη δηλαδή σε σχέση με τον κύριο Λάγκεν. Ε, νομίζω ότι έχουμε αντλήσει πολλά διδάγματα από αυτά που έγιναν για το διοξείδιο του άνθρακα για τα αυτοκίνητα. Είναι κρατεά η αυτοκινητοβιομηχανία και ξαφνιάζει και τον ίδιο τον εαυτό ορισμένε φορές από την ταχύτητα προσαρμογής που έχει και το καλωσορίζουμε αυτό. Και θα έπρεπε να το ενθαρρύνουμε και να δράσουμε κι εμείς αναλόγως ε, όταν θεσπίζουμε διατάξεις για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Μπορούμε και θα έπρεπε να θέσουμε μακροπρόθεσμο στόχο για το 2020 ε, πάνω από τα 120 μικρογραμμάρια όχι μόνο γιατί απέδειξε ε, την ε, ότι είναι, είναι ικανή να προσαρμοστεί η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά ακούω από τον κλάδο ότι χρειάζεται ασφάλεια και μακροπρόθεσμος ε, σχεδιασμός. Οπότε τώρα θα έπρεπε να έχουμε ένα φιλόδοξο αλλά και σαφή στόχο για το 2020. Ας σκεφτούμε και τις ανάγκες ε, των ε, επιχειρήσεών μας ε, που βαρύνονται με αυτό, θα βαρύνονταν με το περιττό άχθος ε, αν επιτρέψουμε να κυκλοφορούν αυτά τα ελαφρά οχήματα χρησιμοποιώντας ε, περισσότερο καύσιμο από ό,τι θα έπρεπε. Μιλήσατε για τη δεκαετή περίοδο, αλλά αυτό που σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε είναι να κυκλοφορούν οχήματα που δεν έχουν καμία φιλοδοξία για την εξοικονόμηση καυσίμου και να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να ε, υπομιστούν το άχθος ε, αυτών των ε, οχημάτων. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Λάγκεν για τον περιορισμό της ταχύτητας. Είναι βέβαια δύσκολο να μιλήσουμε για την εξοικονόμηση του άνθρακα και να την υπολογίσουμε. Βέβαια, μειώνεται η εκπομπή όταν μειώνουμε την ταχύτητα. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί και είναι λογικό. Και ούτως ή άλλως μεγάλες επιχειρήσεις ε, το εφαρμόζουν ήδη σε εθελοντική βάση. Λογικό είναι λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και ε, έχει και άλλα πλεονεκτήματα, την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια ας πούμε. Εμένα μου αρέσουν ε, τα ε, ε, ε, τα ηλεκτρικά οχήματα όχι, και γιατί ξεκίνησαν και στην βορειοανατολική Αγγλία αυτά, αυτές οι σούπερ υπερπιστώσεις επίσης καλοδεχούμενες είναι Με αυτά τα κίνητρα βέβαια για τα ηλεκτροκινούμενα οχήματα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ανεπιθύμητη ε, κατάσταση, δηλαδή παίρνει μια ε, φορολογική ελάφρυνση ο κατασκευαστής ε, επειδή παράγει τέτοια ηλεκτρικά οχήματα, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τα οχήματα που συνεπάγονται μεγάλες εκπομπές και άρα αφήνουμε απ' έξω ένα μεγάλο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, ως προς τις ε, κυρώσεις, ε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το σύστημα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στα 120 μικρογραμμάρια και επίσης ε, χρειάζεται οπωσδήποτε να αντισταθμίσουμε αυτό το ζήτημα των υπερπιστώσεων, των φορολογικών ελαφρύνσεων. Δεν νομίζω επίσης ε, ότι οι κατασκευαστές πρέπει να φέρουν ε, την ευθύνη για το τι συμβαίνει μετά την πώληση του αμαξώματο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μία μεθοδολογία για τα σασί και για τον τρόπο που πρέπει να τα χειριστούμε. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Εμείς πρέπει να βρούμε τη λύση. Η Συνάδελφο Χάλμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Λάγκεν μπορεί να εκπλήσεται από την στάση που έχω κρατήσει. Νομίζω ότι όλοι μας θυμόμαστε τη συζήτηση για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακος, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος στα επιβατικά αυτοκίνητα. Θέλω όμως να σας πενθυμίσω κάτι από αυτή τη συζήτηση, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία ακολούθησε μια συγκεκριμένη πορεία μετά από την συμβιβαστική λύση που κατάφερε να αποσπάσει η αυτοκινητοβιομηχανία για να καθυστερήσει και να αποδυναμώσει την εφαρμογή της πρότασης της Κομισιόν. Μόλις τελειώσαμε λοιπόν τον τριγωνικό διάλογο και αυτό ήταν στη στιγμή που είχε οξυνθεί ιδιαίτερα η οικονομική κρίση στην Ευρώπη όλες οι εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ε, Ευρώπη ξεκινήσαν αυτή την εκστρατεία για τα υπερφιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητά τους. Είδα στι ακριβότερες εφημερίδες και στην τηλεόραση να υπάρχουν ε, διαφημίσεις όλων των εταιριών. Καμία από τις εταιρείες αυτές δεν ήθελε να βρεθεί εκτός νυμφώνος με το να μην έχει να παρουσιάσει ένα αυτοκίνητο που ήταν κάτω από 120 γραμμάρια το χιλιόμετρο. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλουμε να ξαναεπαναληφθεί αυτό το παιχνίδι κύριε Λάγκεν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας, απασχολεί, να μας απασχολήσει ο κίνδυνος η Greenpeace να αποφασίσει ποια θα πρέπει να είναι η νομοθεσία. Είναι πιο ανησυχητικό να υπάρξει επανάληψη του σεναρίου που είδαμε για τα επιβατικά αυτοκίνητα, δηλαδή να παρέμβει η βιομηχανία και να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός ο οποίος αποφασίζεται είναι πόρο απέχων από τις τεχνολογικές δυνατότητες της στιγμής. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι η πλήρης εφαρμογή ενός υποδέστρου στόχου 11 χρόνια, το 2018 δηλαδή, μετά από την πρώτη συζήτηση που κάναμε για το θέμα αυτό το 2007, ένα τέτοιο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να εφαρμοστεί ένας τέτοιος κανονισμός, κύριε Λάγκεν, αυτό δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι αυτό εμπίπτει στα πλαίσια του better regulation είναι περισσότερο business as usual σε ό,τι αφορά την αύξηση της ενεργειακής και ε, περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των οχημάτων και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ λοιπόν. Επίσης ο στόχος του 2020. Και εκεί πάλι θέλετε να αποκλίνετε από αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν. Εσείς λέτε 140 γραμμάρια το 2025 να είναι ο στόχος και αυτό θα σήμαινε ότι τα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα θα, θα του ζητηθεί μονάχα το ίμιση της μείωσης εκπομπών που θα πρέπει να επιτύχουν τα επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι το 2020. Και πάλι αυτό δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή απέτηση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια καλή και φιλόδοξη πρόταση με την οποία εμεί προωθούμε την καινοτομία στην αυτοκίνητο βιομηχανία για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Επίσης και για τα πρόστιμα είναι γνωστή αυτή η συζήτηση. Την είχαμε συζητήσει σε όλα τα επίπεδα με την Κομισιόν για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Τα πρόστιμα έχουν νόημα μόνο αν τα πρόστιμα είναι πιο ακριβά από την εφαρμογή λύσεων οι οποίες είναι τεχνολογικά καινοτόμες. Νομίζω ότι αυτό ήταν η ιδέα της Κομισιόν να είναι υψηλά τα, τα πρόστιμα και δεν καταλαβαίνω γιατί εσείς θέλετε να μειώσετε κύριε Λάγγεν το πρόστιμα προς την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα ήταν πιο λογικό να πείτε ότι δεν θέλετε καθόλου μηχανισμούς κυρώσεων, να μην υπάρχουν καθόλου πρόστιμα παρά μόνο θα ήταν καλύτερο αυτό παρά να προτείνεται ένα επίπεδο προστήμων που ουσιαστικά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η βιομηχανία να πληρώσει τα χρήματα αυτά για να μην εξασφαλίσει την εφαρμογή μέτρων καινοτομία στα αυτοκίνητα. Γενικά για το βιομηχανικό κλάδο στην Ευρώπη της αυτοκίνητοβιομηχανίας νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα όταν η νομοθεσία ζητούσε φιλόδοξες τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομία. Δεν βελτιώνεται η αυτοκινητοβιομηχανία όταν δεν την πιέζεται να είναι πιο αποτελεσματική και να χρησιμοποιεί λιγότερα καύσιμα. Και επίσης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο υποστηρίζεται για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό θα είναι καλύτερο να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση καυσίμων γιατί θα ξανανεύουν οι τιμές του καυσίμου σε παγκόσμιο επίπεδο και επίσης είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και τον στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος που και αυτό το θέμα μετά από την Κοπενχάγη βρίσκεται λιγάκι σε μετεωρισμό. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει εμείς να πιέσουμε για να υπάρξει μια προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών του άνθρωπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ουσιαστικά ήδη από την πρώτη συζήτηση που είχε γίνει γύρω από το θέμα αυτό είχα συμφωνήσει με τις περισσότερες προτάσεις. Τώρα έχει φτάσει η ώρα να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένες αναλύσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα ο οποίος είναι κυρίαρχα οικονομικός θα έλεγα εμπορικός και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα αυτό έχουν σαν βασική ανησυχία το κόστος. Προφανώς και ο όγκος των μεταφερομένων προϊόντων επηρεάζουν ε, τις παραγωγές των ε, κατηγοριών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε αναλυτικότερα πριν πάρουμε κάποιες τελικές αποφάσεις για τον χρονισμό των κυρώσεων οι οποίες θα πρέπει να επιβληθούν. Πρόκειται για κανονισμούς οι οποίοι θα επηρεάσουν άμεσα τον επιχειρηματικό κόσμο και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και δεν θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε ένα σοκ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ήδη βιώνουν οι επιχειρηματίες. Ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων τους και σίγουρα τους ενδιαφέρει βέβαια το να χρησιμοποιούν ένα όχημα το οποίο να κοστίζει λίγο δεν πάβει αυτό να είναι ένα σοβαρό οικονομικό βάρος, μια οικονομική επιβάρυνση και δεν θα πρέπει εμείς με τις διοικητικές μας ρυθμίσεις να καταστήσουμε πιο περίπλοκη την κατάσταση. δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε διαφορετικού τύπου κυρώσεις στα εμπορικά οχήματα από ό,τι στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Νομίζω ότι καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο διοικητικό σύστημα και όχι να εγκαταστήσουμε νέου τύπου μηχανισμούς ε, στα οχήματα αυτά που θα λειτουργούν μόνο και αυστηρά περιοριστικά. Οι αριθμοί στους οποίους θα καταλήξουμε δεν είναι ακόμα αποφασισμένοι. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες των οχημάτων τις οποίες θα καλύψουμε με τους περιορισμούς που θέλουμε να επιβάλλουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Λάγκε ε, για το πώς θα μπορέσουμε να κατανείμουμε καλύτερα την μείωση ε, της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα τα επόμενα χρόνια είναι δυνατόν να έχουμε γρηγορότερες εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας. Είναι επίσης χρήσιμο να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και μία αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας που θα καταναλώνουμε. Η πίεση του κόστους ε, του πετρελαίου και γενικότερα των πρώτων υλών είναι θα έλεγα μία επιπλέον πίεση την οποία υφίστανται οι κατασκευαστές των οχημάτων αυτών. Ο κύριος Ένσο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Μουλτσουμέσκ. Θα ήθελα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκεν για το ε, σχέδιο έκθεσης που υπέβαλε Ξέρουμε όλοι ότι τα ε, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αντιστοιχούν στο 12% του συνόλου του στόλου των οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εφικτό να επιτύχουμε τη μείωση κατά 20% μέχρι το 2020, αναρωτιόμαστε. Μία υπερβολικά ριζοσπαστική νομοθετική ρύθμιση στον κλάδο ενδέχεται να έχει ε, αρνητικό αντίκτυπο και μην ξεχνάτε ότι έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση ο τομέας της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας θα δυσκολευτούν δε ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα οχήματα προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία διότι είναι ένα παραγωγικό μέσο για αυτές τις επιχειρήσεις το ε, επαγγελματικό όχημα. Πιστεύω επίσης ότι θα έπρεπε να παρατείνουμε τις προθεσμίες για την εφαρμογή αυτών των μειώσεων που προτείνει το σχέδιο κανονισμού, ούτω ώστε οι οικονομικοί φορείς να έχουν τον επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους, ώστε να προσαρμόσουν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Ε, οπότε δεν είναι ε, βιώσιμος αυτός ο στόχος ε, των 35 ε, γραμμαρίων. των 135 γραμμαρίων δεν είναι εφικτός. Νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνουμε 120. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο που μίλησε πριν από μένα ε, δεν ε, θα προτείναμε μείωση 5 γραμμαρίων το χρόνο, γιατί δεν μπορούν οι επιχειρήσει σε διάστημα ενός έτους να προσαρμόσουν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Δεν είναι εφικτή αυτή η λύση. Αντίθετα, θα συμφωνήσω με μακροπρόθεσμους στόχους μέχρι το 2025. Ε, τώρα, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα των κυρώσεων και των εισόδων που θα προκύψουν από την επιβολή κυρώσεων. Συμφωνούμε ε, για ε, όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να τηρηθούν οι ποσοστώσεις, αλλά ε, τελικά θα, ένα μέρος του κόστους θα το υπομειστεί ο καταναλωτής. Ευχαριστώ. Nächstes Κύριος Γκρότε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έχω ξαναδεί αυτό το έργο από την ε, συζήτηση της νομοθεσίας για τα ελαφρά οχήματα, όπου υπήρξε μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρόταση με, από τον κύριο Λάγκεν. Εγώ υπήρξα εισηγητής σκιώδης ηγητής για την ε, πρόταση για τα Euro 5 και Euro 6 πρότυπα εκπομπών και βλέπω ότι αυτή η ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί με αρκετά ουδέτερο τρόπο στην αγορά. Και δεν έχει κανένα νόημα να καθυστερήσουμε περισσότερο αυτήν την οδηγία. Αντίθετα με τα επιβατικά οτυχήματα και έχει δίκιο ο κύριος ε, Λάγκεν. Αυτό αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι δεν έχουν επιλογή, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν παρα, παραδόσεις με ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα και δεν έχουν την επιλογή του πώς θα μεταφέρουν αυτά τα αγαθά. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν αυτοκίνητα με συγκεκριμένες διαστάσεις για να κάνουν αυτή την εργασία. Για το θέμα των προστήμων πιστεύω ότι και στην περίπτωση των ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων και στην περίπτωση των ε, επιβατικών αυτοκινήτων δεν δημιουργούμε κυρώσεις κατά των, ε, των κατασκευαστών, ίσα ίσα τους βοηθούμε να προχωρήσουν, να προχωρήσουν σε υψηλή τεχνολογία. Αν υποχρεώνεται λοιπόν ο κατασκευαστής να προβεί σε καινοτομίες, θα πρέπει να έχει και την εγγύηση ότι ένα τέτοιο όριο, αν παραδείγματος χάρη επιβάλλουμε ένα όριο ταχύτητος, ότι αυτό το όριο ταχύτητος πραγματικά θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν αυτό το, το όριο των 120 χιλιόμετρων την ώρα σαν όριο για να υπάρξει μείωση των εκπομπών, αλλά είναι απαραίτητο να ξέρουμε ποια είναι η εξοικονόμηση η οποία θα, θα επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό. Επίσης, σε σχέση με τους κατασκευαστείς του αμαξώματος, του σασί, ποια είναι η ευθύνη αυτών όταν στη συνέχεια παίρνουν το αμάξωμα άλλοι κατασκευαστές και φτιάχνουν μια υπερδομή θα πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Λάγκεν, να μας πει η Κομισιόν με ποιο τρόπο προτείνει να αντιμετωπίσει αυτές τις ειδικέ περιπτώσει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να αφορά μονάχα τον αρχικό κατασκευαστή. Λοιπόν, ο ενδιάμεσος στόχος των 175 γραμμαρίων είναι εφικτός να επιτευχθεί το 2014. Τι γίνεται με το μακροπρόθεσμο στόχο. Απαιτεί ένα τεχνολογικό άλμα, μια αλλαγή τεχνολογιών και πιστεύω ότι με τα τωρινά δεδομένα ο στόχος του 135 γραμμαρίων δεν είναι εφικτός. Έχουμε χρόνο όμως. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουμε βάλει το στόχο των 120 μέχρι το 2020 και νομίζω θα ήταν σωστό να βάλουμε κάποιους φιλόδοξους στόχους και σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε διαφορές μεταξύ σας για το χρονικό ορίζοντα και πώς θα υπάρξει η σταδιακή εφαρμογή αυτού του στόχου των 135 γραμματείων. Πιστεύω ότι από την έποψη της βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό το στόχο γιατί αποδυναμώσουμε αυτό το στόχο δεν θα μπορούν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί δεν θα έχουν τα αυτοκίνητα εχμής. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε με την, ε, να παραμείνουμε στο επίπεδο της πρότασης Κομισιόν και για τους, ε, τα οχήματα με πολλαπλούς κατασκευαστές θα πρέπει να περιμένουμε να μας πει η Κομισιόν με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και να δούμε λοιπόν πώς για τα ελαφρά οχήματα θα επιτύχουμε τους στόχους που είχε θέσει ο κύριος Σακώνη στην εκθεσή του. Δεν πρέπει να δεχτούμε λοιπόν την αποδυνάμωση των στόχων από τον κύριο Λάγκερ. Νομίζω ότι εμείς με τον τρόπο αυτό δεν βοηθούμε τη βιομηχανία, απλώς ε, καθυστερούμε την προσαρμογή της. Ξέρω ότι ο κύριος ε, Λάγκεν θα ακολουθήσει μια διαφορετική άποψη και για τις ε, υπερπιστώσεις, τα super credits, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα, δεν πρέπει να τα αποδυναμώσουμε. Μιλάμε για ένα τεχνολογικό άλμα. Χρειάζεται να ευνοήσουμε τη νέα τεχνολογία και επομένως θα πρέπει να επιβραβεύσουμε και τους κατασκευαστές οι οποίοι χρησιμοποιούν μια νέα τεχνολογία, κάτι το οποίο πρέπει να το διατυπώσουμε με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν και να είναι πρωτοπόροι. Επομένως αυτά τα super credits, αυτές οι πρόσθετες πιστώσεις βοηθούν τη βιομηχανία. Και πρέπει επομένως και οι βιομηχανίες να τύχουν αμοιβή για την τεχνολογική τους αυτή πρόοδο. Ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα υποστηρίξω τις προτάσεις του συναδέλφου Λάγκεν γιατί δείχνει ιδιαίτερη σύνοση και έτσι πρέπει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα μέτρα αυτά απορρέουν από μια συμβαστική πολιτική λύση ε, που αποφασίσαμε στα τέλη του 2008, τρεις φορές 20, ε, δηλαδή μείωση 20-20-20 μέχρι το 2020. Βέβαια, ε, στην Κοπενχάγη δεν αποφασίστηκε καμία οικουμενική συνένεση, εν αναμονή μιας παγκόσμιας συμφωνίας, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως το παρελθόν και να επιβάλλουμε δηλαδή περιορισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία ενώ οι ανταγωνιστές τους στη διεθνή σκηνή δεν ε, συμμορφώνται με τους ίδιους περιορισμούς. Γι' αυτό χρειάζεται σύνεση τουλάχιστον ε, για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Ε, είπαμε προηγουμένω ότι είναι ισχυρή η αυτοκινητοβιομηχανία. Ναι, αλλά προσοχή, αν υπολογίσουμε τις, τις ε, κυρώσεις, οι υπολογισμοί ε, οδηγούν γρήγορα σε ένα-δύο χρόνια κερδών ε, για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Προσοχή! Τι θα βάλουμε στους ώμους ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας με αυτές τις κυρώσεις. Δεν μπορεί να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κατασκευαστές που θέλουν να κατασκευάσουν οχήματα 150 γραμμαρίων στην Ευρώπη που πρόκειται να εξαχθούν ε, σε χώρες όπου δεν ισχύουν οι ίδιες αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις. Είδω κάποιες παρατηρήσεις για να υποστηρίξω τις προτάσεις του συναδέλφου Λάγκεν. Ευχαριστούμε. Μήπως θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Λάγκεν για το σχέδιο έκθεσης και ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές που πήραν το λόγο σήμερα. Για να δούμε ποια είναι η συνολική εικόνα. Πέρσι τον Οκτώβρη οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν για κάποια συμπεράσματα για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ φιλόδοξο ο στόχο, αλλά χρειαζόμαστε και τι αντίστοιχε πολιτικέ ε, για να τα εφαρμόσουμε αυτά σαφέστατα. Αν δείτε τι προβολέ για το μέλλον, ε, ε μεγενθύνεται το τομέα ε, των μεταφορών, κυρίω όταν μιλάμε για μεταφορέ εμπορευμάτων και από εκεί απορρίνουμε μεγαλύτερε εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου. Οπότε, ελοχεύει ο εξή κίνδυνο. Αν δεν δράσουμε τώρα και αν δεν λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα, ε, να τελικά οι μεταφορέ να δίνουν το 100% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σήμερα μέσα από τις πολιτικές μας. Αυτή είναι η συνολική εικόνα και πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσαν επανειλημμένα οι βουλευτές. Πρώτον, το θέμα του κόστους. Για όσους διάβασαν ε, την ε, μελέτη αντικτύπου και την ανάλυση θα δουν ότι είναι ουδέτερη ε, ως προς το κόστος. Ε, δηλαδή μέχρι το 2020 ο στόχος του 135 γραμμαρίων δίνει πλεονέκτημα γιατί η εξοικονόμηση του καυσίμου αντισταθμίζει το επιπρόσθετο κόστος και τελικά είναι ωφέλιμο για τον καταναλωτή και επίσης θα μειωθούν οι εκπομπές το οποίο είναι και καλό για την κοινωνία. Αυτό προκύπτει από την μελέτη αντικτύπου της Επιτροπής ε, και αυτά που ακούστηκαν ε, ότι θα ε, αυξηθεί το κόστος δεν νομίζω ότι προκύπτει αυτό από την ανάλυση. Τώρα το θέμα των ακυρώσεων. Γιατί τα 120 ευρώ αναγραμμάριο. Μα 95 ήταν για τα αυτοκίνητα και αυτό ήταν το οριακό κόστος και αυτό λέμε στην αξιολόγηση αντικτύπου. Οπότε οι κατασκευαστές θα επιλέξουν να κάνουν την οριακή προσαρμογή αντί να ε, τους επιβληθεί το πρόστιμο. Αυτή, αυτό είναι το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κάτι άλλο που άκουσα επανειλημμένα είναι το θέμα των ε, μηχανισμών ελέγχου της ταχύτητας είναι, παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτό το μέτρο και ούτω ή άλλω υπάρχουν ταχύμετρα μέσα στα φορτηγά ε, και δεν μιλάμε για εθνικά ταχύμετρα. Ε, ε, δεν ε, παρεμβαίνουμε δηλαδή στην εθνική κυριαρχία. Θα μειώσουμε όμω ε, αν γίνει αυτό σε εθελοντική βάση, την κατανάλωση του καυσίμου και άρα και τι εκπομπέ ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Θα έχουμε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και ε, θα καλύψουμε και άλλε τέτοιε συναφείς πτυχέ. Τώρα, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε πολλά στάδια. Άκουσα πολλά σχόλια και εδώ είχαμε υποβάλει ανεπίσημη πρόταση προς το Συμβούλιο και προς την Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε συμφωνήσει για το μέλλον, δηλαδή πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό το θέμα των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται ε, σε πολλά στάδια. Και ε, συμπεριλάβατε τις παρατηρήσεις μας ε, στο έγγραφο εργασίας σας για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οπότε θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Γκρότε. Ε, για τα υπόλοιπα ζητήματα ε, εμένουμε στην πρότασή μας. Ε, το, το, ε, ο στόχος των 175 μέχρι το 2060 είναι εφικτός στόχος και τα 100 μέχρι το 2016 είναι ένας εφικτός στόχος και χρειάζονται βέβαια τεχνολογικές ε, προσαρμογές, αλλά αν γίνουν ε, είναι υλοποιήσιμο ο στόχος. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει καινοτομία στον ε, τομέα. Μίλησαν πολύ για ανταγωνιστικότητα. Ο κύριο Σοντή, παραδείγματο χάρη, είπε ότι δεν θα πρέπει να αποφύγουμε να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα με το επιπρόσθετο κόστος. Μα το αντίθετο συμβαίνει γιατί ε, σπρώχνουμε την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να καινοτομήσει τώρα, ώστε μέχρι το 2020 να έχει πιο αποδοτικά οχήματα ε, που ε, που υπάρχουν ήδη στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία. Δηλαδή θέμα χρόνου είναι για να βρεθούμε ε, στην, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε 135 γραμμάρια μέχρι το 2020 και 160 μέχρι το 2016. Ε, τώρα πρέπει να περάσουμε το σωστό μήνυμα στην αυτοκινητοβιομηχανία για τα ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτό αυτή η πρόοδος πρέπει να σημειωθεί και θα, θα χρησιμοποιήσουμε τις κρατικές προμήθειες στο δημόσιο τομέα, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση. Αυτά τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν σε αστικές περιοχές ε, για τα χειδρομικές υπηρεσίες, ε, για τις παραδόσεις αγαθών κτλ. Οπότε ε, η πράσινη πολιτική στις κρατικές προμήθειες είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Συμπερασματικά θα, ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα σχόλιά του και με αυτό το νομοθέτημα θα δώσουμε και την ασφάλεια ως προς τον πραγματισμό που χρειάζεται η αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, και μένουμε στην πρότασή μας. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Είχα δει ένα έγγραφο πρόσφατα το οποίο ασχολιόταν με το θέμα αν πρέπει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο πρόδρομοι των αλλαγών για την κλιματική αλλαγή και φανταζόμαι και σε άλλα θέματα. Ίσως δεν είναι τώρα ερώτημα για το συγκεκριμένο έγγραφο, αλλά νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα προβληματική να δούμε κατά πόσο πράγματι μας ενδιαφέρει να παίξουμε αυτό το ρόλο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λάγκε, ναι. Θα ξεκινήσω με την παρατήρηση του εκπροσώπου της Κομισιόν. Είναι σαφές ότι έχουμε προτείνει μέχρι το 2050 να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακος κατά 80-90% και αυτό δείχνει ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ε, σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόμα και αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα μειώσει κατά 100% τις εκπομπές μέχρι το 2050, και δεν θα εκπέμπαμε τίποτα. Οι Κινέζοι δεν θα το δεχόντουσαν γιατί αυτοί έχουν μια άλλη ιδεολογία, έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να έχουμε αποφάσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την διατήρηση της ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρώπης και δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις οι οποίες θέλουν 40 χρόνια για να εφαρμοστούν στην πράξη. Για μένα λοιπόν η Κομισιόν δεν μας προσφέρει τίποτα με αυτά που λέει για την για τις πράσινες προμήθειες σε επίπεδο οχημάτων. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι δεν είναι αυτή ο νομοθέτης, αλλά είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και πρέπει να ληφθεί από αυτό υπόψη στις αποφάσεις μας για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τα ελαφρά αυτοκίνητα. Υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι εδώ οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη ότι θα πρέπει να κινηθούμε με προσοχή, ότι θα πρέπει να ελέγξουμε καταρχήν αν η στόχη είναι επιτεύξιμη και εφικτή και τέθη το ερώτημα του γιατί θέλουμε να παρατείνουμε την, ε, τον χρονικό τον χρονικό οριζόντα της επίτευξης του στόχου για τα 140 γραμμάρια. Νομίζω ότι πάντα το όριο αυτό, η βάση υπολογισμού αφορά το συνολικό στόλο αυτοκινήτων που παράγει ένας ε, κατασκευαστής, αν κάθε χρόνο αλλάζει ένα μοντέλο από τα πολλά, αυτός ο στόχος είναι επιτευτό, επιτεύξιμος. Μπορούμε να έχουμε διαφορές σε σχέση με, το, με, την, ε, με τα συγκεκριμένα αριθματικά στοιχεία, αλλά εγώ πιστεύω το ότι τα 135 γραμμάρια το 2020 είναι ανέφικτο. Και κυρία Χάρμς, είπε ότι δεν πρόκειται για την Greenpeace που προσπαθεί να περάσει αυτή την άποψη, αλλά ουσιαστικά η κυρία Χάρμς ανέφερε τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία είχε διατυπώσει η ίδια η Greenpeace. Μίλησε για τα 11 χρόνια που χρειάζεται η εφαρμογή, 2007 με 2018. Εμείς δεν μιλάμε για 11 χρόνια, δεν ξεκινάει το 2007. Το 2011 θα ξεκινήσει αυτή η νομοθεσία σε εφαρμογή. Αλλά λέει επακριβώ χαλκομανία αυτά τα οποία λέει η Greenpeace. Ακριβώς αυτό λέτε. Αυτό θέλω να σας πω. Ακριβώς τα τρία σημεία τα οποία είπε η Greenpeace. Τα έχω εδώ πέρα να σας τα δείξω. Και απλώς ανταποκρίνεστε απόλυτα σε αυτά τα οποία είπε η Greenpeace. Εγώ είμαι έτοιμος να προχωρήσω σε διάλογο αλλά νομίζω ότι τα δικά μου επιχειρήματα πρέπει να τα αντικρούσετε με ουσιαστικά επιχειρήματα. Άκουσα επίση την πρόταση ότι θέλουμε να έχουμε φιλόδοξους στόχους από τον κύριο Οντί, Γκρότε, Μπιρέλη, Χολτ κτλ. τα Χαίρομαι για τις προτάσεις αυτές που παρουσίασαν. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για επαγγελματικά αυτοκίνητα που έχουν να κάνουν με μικρούς παραγωγούς. Υπήρξε <clears throat> μια μεγάλη πρόοδος στην τεχνολογία αυτών των αυτοκίνητων και το γεγονός ότι τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα φτάνουν τα 6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, αυτό δείχνει την πρόοδο της τεχνολογίας. Η τεχνολογία πρέπει να μείνει στα πλαίσια του εφικτού. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μπορεί η αυτοκινητοβιομηχανία να αλλάξει άρδιν την αντιμετώπιση της. Η αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να λειτουργήσει με εθελοντική βάση αυτή η ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτό δεν λειτουργήσε. Πρέπει να έχουμε νομοθεσία, αλλά είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες των κατασκευαστών ε, μικρών επαγγελματικών ε, οχημάτων και επομένως είναι απαραίτητο να καταλήξουμε στις απαραίτητες λύσεις για να φτάσουμε και σε ένα συμβιβασμό με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν. Εγώ δεν νομίζω ότι με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε τα θέματα αυτά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θέλω να κάνω απόλυτα σαφές ότι από τη δική μας πλευρά οι στόχοι μείωση του διοξιδίου του άνθρακο, που είναι το υπόβαθρο για αυτή την νομοθετική πρόταση θα είναι αυτοί που έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα άλλο αλλά να ενσωματώνει τις προτάσεις αυτές τις προτάσεις αυτές που έχουν ουσιαστικά αποφασίσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το 2007 υπό την ηγεσία και την παγέτα της κυρίας Μέρκελ. Και αυτά συμφωνήθηκαν στο Νταμ και δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτή τη στοχοθεσία μετά την Κοπενχάγη. Εγώ θα ήλπιζα τώρα να υπάρχουν ε, προτάσεις από την κυρία Χέντεγκαρτ και από την Κομισιόν να υπάρξουν πραγματικά συγκεκριμένε προτάσει και όχι απλώ προτάσει οι οποίε προχωρούνται από του κόλπου τη βιομηχανία. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρο, δεν θέλω να κάνω μία. Αυτή δεν ήταν διαδικαστική παρέμβαση, κυρία Χάμ, αλλά όλα αυτά είναι ζητήματα πολιτική αξιολόγηση. Ο καθένα έχει το δικαίωμα, ο κάθε συνάδελφο έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτική στοχοθεσία και μπορεί να διαφυσβητεί τις απόψεις των άλλων και τις θέσεις των άλλων. Έχουμε πολλές φορές την ανάγκη να αναθεωρήσουμε τους στόχους, τους πολιτικούς που θέτουμε στην πορεία. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι απόλυτα κύριε Λάγκεν θεμητό να δέχεται κανείς και να μεταφέρει προτάσεις ενός φορέα όπως η Greenpeace. Και εξάλλου υπάρχει και αντίστροφα το δικαίωμα. Μπορεί κάποιος από μια άλλη πολιτική ομάδα να μεταφέρει προτάσεις αυτοκινητοβιομηχανίας και αυτό είναι εξίσου εφικτό και είναι εξίσου θεμητό. Αν λοιπόν και οι δύο πλευρές πράττουν ούτως, έχουμε μια καλή αντιπαράθεση απόψεων και νομίζω και η συζήτησή σας συνέβαλε σε αυτό το στόχο. Κύριε Λάγκεν, αλλά όχι διαδικαστικά σας παρακαλώ. Εγώ δέχομαι απόλυτα αυτό το οποίο είπατε σε σχέση με την εκπροσώπηση άλλων φορέων. Απλώς έκανα αυτήν <clears throat> την... Ε, έκανα την παρατήρηση γιατί η κυρία Χάμς είπε ότι δεν είχε καμία σχέση η πρότασή τη με αυτήν τη γκρίπη. Εντάξει, έχει διαλευκανθεί αυτό το θέμα, αλλά στο μέλλον μπορεί ο καθένα χωρί ψόγο να φέρνει προτάσει από οποιοδήποτε φορέα. Λοιπόν, διακο... Ε, διακοπή ως τις 3 ώρα και θα επανέλθουμε. Α, για την καταληκτική ημερομηνία, συγγνώμη. Ζητήθηκε να καθυστερήσει, το έλεγξε η γραμματεία, δεν είναι τόσο εύκολο. Θα προσπαθήσει η γραμματεία. Το πρόβλημα είναι ότι ο... οι υπηρεσίε μετάφρασης είπαν ότι το αργότερο στις 4 ή στις 6 Μαΐου να έχουν έλθει τα έγγραφα γιατί αλλιώς θα καθυστερήσει λόγω των διακοπών. Θα προσπαθήσει λοιπόν η γραμματεία να φτάσουμε στις 7. Λοιπόν, δεν είναι αποφασισμένη η προθεσμία, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα. Εντάξει. Αν γίνεται φυσικά θα το καθυστερήσουμε. σε μια άλλη επιτροπή είδα ότι παρά τις διακοπές του Πάσχα κράτησε δύο εβδομάδες μονάχα η μετάφραση των τροπολογιών. Αυτό έθεσε του συναδέλφου σε τεράστια πίεση, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε τίποτα. Αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, λέει ο πρόεδρο.